Uh, um, Συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε. Βέβαια το ακροτήριο είναι υψηλής ποιότητας, αλλά χαμηλής ε, πυκνότητας, θα μπορώ να πω έτσι. Ε, οπωσδήποτε όλοι θα ακούσουν με πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχετε να μας πείτε. Θα περιμένω να, ακούσω, να έρθει ο κ. Στάλι εδώ για να κάνω κάποιες ανακοινώσει. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίως υπεύθυνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ήβεν και Σάτη γιατί ε, έγινε χθες μια πολύ καλή διαπραγματευτή συνεδρίαση και πλησιάζουμε θα έλεγα την ε, συμφωνία. Πολύ καλό παράδειγμα ε, ομαδικής εργασίας από το ΒΕΠΑ και το ΜΑΤΑ Χθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κανονίσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα πλευράς της εσωτερικής αγοράς Το θέμα ξέρω ότι θα συζητηθεί και μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για τις ε, υπηρεσίες το εξετάσαμε λίγο και θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται τώρα και οπωσδήποτε εμείς είμαστε υπέρ της υποστήριξης αυτού του σχέδιου. Λοιπόν είναι ψυχνά εδώ. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο και να μας κάνετε την παρουσίαση και μετά ο καθένας μπορεί να υποβάλει μια ερώτηση. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Um, we thought that just giving you presentations on facts... Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αν σας δώσουμε απλώς πληροφορίες γενικές θα ήταν πολύ εμ, δυσνόητο. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να σας ε, δώσουμε δυνατότητα να περάσετε το σύστημα σαν να ήσασταν κάποιος που εργάζεται, ας πούμε ένας Γάλλος αρχιτέκτονας που μετακομπή, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε υποβάλει τα έγγραφά του στις αρχές και θέλει να εγκριθούν τα διπλώματά του και οι επαγγελματικές του ε, τα επαγγελματικά του έγγραφα. ίσως δεν ξέρει κατά πόσον ε, αυτός μάλλον που είναι στο γραφείο στο Ενωμένο Βασίλειο δεν ξέρει αυτό το πιστοποιητικό, αυτό το δίπλωμα που του δίνουν. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που θέλουν ίσως να εξετάσουν που του δώσουν το πράσινο φως. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να πάνε στον πολύγλω... στην πολύγλωση ιστοσελίδα του IMI για να πάρουν τους προφέρειες. Δεν θέλουν δηλαδή ειδικό software, ειδικό λογισμικό στους υπολογιστές σας, αλλά μπορούν να το κάνουν μέσα του ε, υπολογιστή τους. Μετά έχει, υπάρχει αυτή η σελίδα για να εγγραφούν όνομα του χρήστη, ε, προσωπικό κωδικό και έναν κωδικό ασφαλείας όπως αυτός που χρησιμοποιείται για τις τράπεζες. Αυτό της ασφαλή δυνατότητα είναι μόνο για τους ε, εγκεκριμένους χρήστες των αρμοδίων ε, αρχών. Είναι πάρα πολύ ασφαλή λοιπόν αυτά τα στοιχεία που ανταλλάσσονται. Μετά, ε, οι αρχές για την καταγραφή των αρχιτεκτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγουν στη γλώσσα τους την σελίδα IMI. Ο καθένας μπορεί να έχει τις πληροφορίες στη δική του γλώσσα, όπως σας είπα. Και βέβαια υπάρχει έτσι ένα καλωσόρισμα στην αρχή και μετά η αρμόδια αρχή έχει όλα τα διαθέσεις, διαθέσιμες ε, πράξεις ε, για τον χρήστη ανάλογα με το προφίλ του ε, γιατί καμιά φορά υπάρχουν περισσότερες, λιγότερες πληροφορίες αλλά αυτό που κάνει το IMI είναι να στείλει ε, το αίτημα αυτό σε άλλες αρμόδιες ε, αρχές. Δηλαδή, εάν η αρμόδια αρχή ε, μπορεί να υποβάλει ερωτήσει για πολλούς νομικούς τομείς, περισσότερους του ενός δηλαδή, γίνεται μια επιλογή για, τις, για τις επαγγελματίες, για τις υπηρεσίες, για τους εργάτες πρόσφατα και προσεγώς θα έχουμε και για τα δικαιώματα των ασθενών. Και λέγεται ποιος θα πρέπει, με ποιον θα πρέπει να έρθουν σε επαφή στη Γαλλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ορισμένες χώρες είναι αποκεντρωμένες. Ας πούμε όμως ότι οι αρχές ε, του Ηνωμένου δεν ξέρουν ποιο πρέπει να έρθουν ε, σε επαφή μπαίνουν λοιπόν στο IMI και ψάχνουν. Το πρώτο κριτήριο είναι η χώρα ή να πούνε αρχιτέκτονας ή και να γράψουν και ένα ελεύθερο, ελεύθερο ένα κείμενο αν αυτό το επάγγελμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα χαρακτηρισμένο. Άμα γράψετε Γαλλία και αρχιτέκτονας. Έχετε ένα κατάλογο 28 αρχών στην Γαλλία που ασχολούνται με αρχιτέκτονες. Όπως βλέπετε σε αυτό τη διαφάνεια ή στο χαρτί που έχετε μπροστά σας γιατί δεν φαίνεται έτσι από μακριά, είναι αποκεντρωμένες οι αρχές στη Γαλλία αυτές και βρίσκονται στο τοπικό επίπεδο. Ας πούμε ότι είναι από την Άνω Νορμανδία ο αρχιτέκτος αυτός και εκεί έχει πάρει και όλα τα διπλώματα. Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο περνάει στις ε, τοπικές αρχές για την Άνω Νορμανδία και εκεί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες με διάφορα στοιχεία για την επαφή που έχουν έχει εγγράψει η εν λόγω αρχή. Ας πούμε στη, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται να τηλεφωνήσουν πρέπει να μιλάνε γαλλικά γιατί οι χρήστες από την άλλη μεριά μιλάνε μόνο γαλλικά και όχι αγγλικά τους χάρη και το ίδιο μπορούν να ελέγξουν ότι αυτή είναι η αρχή πραγματικά που ασχολείται με την αναγνώριση uh, των προσόντων και διπλωμάτων. Και με τι άλλο ασχολούνται. Όλα αυτά είναι βάση κάποιων ε, λέξεων κλειδί που έχουν επιλεχθεί από την ε, υπηρεσία αυτή. Όταν επιλεγεί αυτή η αρχή, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να προετοιμάσει την αίτηση για πληροφορίες. Υπάρχει εκεί ένα κουτάκι που λέγεται μέχρι πότε χρειάζεται την απάντηση. Μέσα στο IMI δεν υπάρχουν επίσημες προθεσμίες, τυπικές προθεσμίες, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα τέτοιο, αλλά μπορούν οι αρχές να πούνε, ας πούμε, εγώ χρειάζομαι την απάντηση στις πέντε μέρες. Και η εμπειρία δείχνει ότι στις περισσότερες ε, περιπτώσεις θα ληφθεί υπόψη αυτό από την άλλη πλευρά και θα εργαστούν γλίγορα. Και θα συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του εν λόγω αρχιτέκτονα, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλικία κλπ. Και ό,τι άλλο Και μετά από μια μακρά σειρά ερωτήσεων που έχουν προοριστεί και μεταφραστεί, μπορεί να κάνει κανένας μια επιλογή ο κατάλογος αυτός είναι χωρισμένο σε ομάδες για να μπορεί πιο εύκολα να το καταλάβει κανένα. Παραδείγματος εδώ στην οθόνη βλέπετε ερωτήσεις που είναι κατά πόσον μπορείτε εσείς να εκδώσετε ένα έγγραφο επίσημα όσον αφορά την πνευματική υγεία του λεγόμενου François Λεγκρό εδώ. Ίσως για αρχιτέκτονες αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, για άλλα επαγγέλματα ίσως είναι σημαντικό. UK authority clicks the questions to ask. Λοιπόν, επιλέγει κανένα τι ερωτήσει θέλει να ρωτήσει, μπορεί και να συμπληρώσει με δικά του σχόλια και επίσης θα μπορέσει να προσαρτήσει έγγραφα και να ε, υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα εν λόγω έγγραφα και υπάρχει και ένα κουτί εδώ, μια δυνατότητα για ελεύθερο ανοιχτό κείμενο. Και βλέπετε ότι αναφέρεται επίσης σε ποια γλώσσα μπορούν να διαβάσουν τις πληροφορίες. Και αυτή η αρχή έχει γράψει ότι μπορεί να διαβάσει και στα γαλλικά και στα αγγλικά. είναι οι δυνατότητες δηλαδή. Εκτός αυτού μέχρι πρόσφατα ε, είμαστε συνδεδεμένοι με το μηχανικό σύστημα μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν σε θέση να μεταφράζει τα σχόλια στην εκάστοτε γλώσσα, αλλά κατόπιν μια απόφαση του δικαστηρίου του περασμένου έτους, αναγκαστήκαμε να αποσυνδεθούμε από το σύστημα αυτό. Και ελπίζουμε ότι ο διάδοχο του συστήματος αυτού θα είναι έτοιμος του χρόνου, γιατί πολλοί από τους χρήστες μας το ζητήσαν και φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εκτός από τις προμεταφρασμένες ερωτήσεις, να μπορεί να μεταφραστεί το ελεύθερο κείμενο. Λοιπόν, τι γίνεται από την άλλη μεριά. Το Γαλλικό Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων παίρνει ε, την ειδοποίηση ότι κάποιος ζητάει πληροφορίες. Και καταρχήν παίρνουν μια περίληψη περί τίνου πρόκειται. Και βάσει της περίληψης αυτής μπορεί να ε, συμφωνήσουν να δεχθούν το αίτημα αυτό και να το επεξεργαστούν ή να το στείλουν σε κάποια άλλη αρχή. Δηλαδή πριν δεχθούν το αίτημα η αρχή αυτή δεν βλέπει τα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω επαγγελματία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σεβαστούμε τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν ανοίξει αυτό το αίτημα για πληροφορίες μπορούν επίσης να περάσουν σε έναν προκαθορισμένο κατάλογο απαντήσεων. Οι απαντήσεις αυτές είναι στα γαλλικά και μπορούν να τα δουν και μπορούν να έχουν και σχόλια ελεύθερα. Το σύστημα καταδεικνύει πάλι ποιε είναι οι γλώσσες που μπορούν να διαβάσουν οι αρχέ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίπτωση. Το Γαλλικό Περιφερειακό Συμβούλιο απαντά στις Βρετανικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται με ένα email, μπαίνουν στο σύστημα, εξετάζουν την απάντηση και βάσει την απάντηση ή τη δέχονται ή ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, αν αυτές που έλαβαν δεν τους αρκούν. Εάν γίνει δεχτή η απάντηση, κλείνει το αίτημα αυτό και είναι σημαντικό αυτό γιατί για την προστασία των δεδομένων ε, πρέπει έξι μήνες μετά που κλείνει το, το αίτημα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα να διαγραφούν από το σύστημα. Αυτά με δύο λόγια. Η βασική ροή των πληροφοριών και ο τρόπος της του IMI. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα που λέγεται alert προειδοποίηση, δηλαδή όπως ξέρετε στην ε, οδηγία για τις ε, υπηρεσίες υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν αν υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα από κάπου που προσφέρει υπηρεσίες ε, και που απειλεί τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, αν κάποιο διαδρά διασυνοριακά, δεν μπορεί, αρκούν να ληφθούν μέτρα στη μία χώρα και μπορεί να αποσταλεί λοιπόν ε, μία προειδοποίηση. Και με την ίδια αρχική σελίδα που σας έδειξα στην αρχή, μπορεί να αποσταλεί αυτό το μήνυμα προειδοποίησης ε, κρούσης του κόδωνα του κινδύνου, αν θέλετε, και υπάρχει εδώ ένας καταλόγος κριτηρίων γιατί δεν θέλουμε να αποστέλλεται ε, μια τέτοια προειδοποίηση αν δεν είναι πραγματικός ο κίνδυνος. Υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων κατά πόσο αυτό είναι ένα κίνδυνος για την υγεία ή για το περιβάλλον, εάν έχει διασυνοριακό πραγματικά χαρακτήρα, εάν σχετίζεται με την προσφορά μιας υπηρεσίας και μετά μπορούν να δημιουργήσουν, να απαντήσουν θετικά σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορούν να δημιουργήσουν αυτό την ε, προειδοποίηση που δίνει τις τα λεπτομέρειες εκείνου που προσφέρει τις υπηρεσίες και του προβλήματος που παρουσιάζεται. Η αποστέλουσα αρχή επιλέγει τα κράτη-μέλη προς τα οποία θέλουν να στείλουν την προειδοποίηση αυτή, που θα πρέπει να είναι κατά τον περιοριστική. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλοι που πρέπει να πάρουν την προειδοποίηση αυτή την παίρνουν και όταν αποσταλεί αυτή η προειδοποίηση μπορούν αυτοί στους οποίους έχει αποστολή να πάρουν ένα email και να εξετάσουν το περιεχόμενο του συστήματος. Και μπορεί μέσα στα πλαίσια του IMI να ανταλλάξουν πληροφορίες εκείνοι που στέλνουν την προειδοποίηση εκείνη που λαμβάνουν και να ζητηθούν περισυμπλωματικές πληροφορίες ενδεχομένω για να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όταν ληφθούν τα μέτρα αυτά και δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος, κλείνει η προειδοποίηση αυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους πάλι προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γιατί εφόσον δεν υπάρχει ο κίνδυνος, τα προσωπικά στοιχεία μέσα στο σύστημα θα διαγραφούν μετά ένα χρονικό ε, όριο. Αυτό είναι το σύστημα έχουμε και ένα άλλο σύστημα που λέγεται registers ε, και αυτή η κατάλογη είναι 800 περίπου στα κράτη-μέλη και επίσης ε, σκοπεύουμε να προετοιμάσουμε κάτι για την κοινοποίηση των εθνικών κανόνων. Εργαζόμαστε λοιπόν για να διευρυνθεί περισσότερο το IMI. Θα κλείσω εδώ, αλλά με ευχαρίστηση θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε για να καταλάβουμε το εύρος και των, των μέσων αυτών που έχουν οι αρμόδιες αρχές στα χέρια τους. Διάφορα έχουν ζητήσει την ερωτήση, αλλά θα δώσω στον αδέρφο στη δυνατότητα να υποβάλουν πρώτα εκείνες τις ερωτήσεις και μετά θα υποβάλω τις δικές μου. Θα ήθελε κάποιος να αρχίσει. Όσο το σκέφτεστε, θα μπορέσω να παρουσιάσω τις δικές μου. Θα μπορούσα ως πρόεδρος ε, να σε μεταλλευτώ τη δυνατότητα να θέσω λίγες φορές το κάνω πρώτο στις ερωτήσεις. Δύο πράγματα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σχετίζονται μεταξύ τους. Πρώτον, έχετε κάποια ένδειξη για το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα κλίμακα μέγεθος διασυνοριακής δραστηριότητας. Δηλαδή υπάρχουν αρχές που το χρησιμοποιούν περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις, τα alerts. Ξέρετε ότι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που μας ανησυχεί ιδιαίτερα έχει να κάνει με την ε, ασφάλεια των ασθενών και το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό των γιατρών για κάποιες θεραπευτικές αγωγές. Υπάρχει και το θέμα όμως προστασίας των δεδομένων που μπαίνει στη μέση και γνωρίζετε φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης από ό,τι φαίνεται σε πληροφορίες για ειδικού ε, γιατρού, ε, ειδικευμένου γιατρού σε κάποιου τομεί. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα όταν οι γιατροί αυτοί μετακινούνται σε μια άλλη χώρα και οι αρμόδιε αρχέ δεν δίδουν κάποιε σημαντικέ πληροφορίε για κάποιους γιατρούς και ενδεχόμενα προβλήματα που είχαν στο ιστορικό αντιμετώπιση, θεραπευτική αντιμετώπιση κάποιων ασθενών. Θα μπορούσε ίσως λοιπόν, επειδή έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια συστήματα και μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει μια προειδοποίηση, να σημάνει σε ένα γερμό. Ε, τι γίνεται ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Βερσιά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βερνιό, κύριε Πρόεδρε, τα τρία τέταρτα των ερωτήσεών μου τα θέσατε εσείς, οπότε θα είμαι πολύ σύντομη. Ξέρετε ότι με μια ομάδα εξετάζουμε το θέμα της εναρμόνισης ε, των επαγγελματικών προσόντων και εγώ για την Ευρώπη του αύριο θα ήθελα να υπάρχει ε, μια επαγγελματική κάρτα, ένα επισκεπτήριο επαγγελματικό, αν θέλετε. Πώς μπορεί λοιπόν να, να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ενημέρωση για την κινητικότητα και των γιατρών αλλά και άλλων μηχανικών, αρχιτεκτών κτλ μπορεί γρήγορα να λειτουργήσει αυτό το σύστημα για να μπορούμε πραγματικά επίσης γρήγορα να οργανώσουμε την κινητικότητα σε κάθε ασφάλεια για τους πολίτες και εντάξει για τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα αλλά μετά γενικότερα για τους πολίτες και μέσα σε πιο χρονικό ορίζοντα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? και μετά η Χάιντι Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά με ενθουσιάζει η εξέλιξη του συστήματος αυτού. Ε, θυμάμαι τις πρώτες παρουσιάσεις ε, που ήταν έτσι κάπως χοντροκομμένες και γινόταν μια αναζήτηση πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Θα το τονίσω αυτό. Και αυτό επιλύθηκε με τον τρόπο ότι δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει κανένας αυτό στον υπολογιστή του, γιατί είχαμε το πρόβλημα το πώς θα λειτουργήσει, μια που υπάρχουν διαφορετικά συστήματα υπολογιστών κλπ. Όλα αυτά επιλύθηκαν. Πάρα πολύ καλό μου φαίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Με τον τρόπο, νέο τρόπο αυτό λειτουργίας ξεπεράστηκε και ένα άλλο πρόβλημα ότι υπήρχε το ερώτημα δηλαδή για ποια επαγγέλματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Τώρα από ό,τι κατάλαβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τομείς χωρίς περιορισμούς. Πολύ σημαντικό αυτό. αν σας κατάλαβα καλά, μπορείτε να μου απαντήσετε, μάλλον με ναι θα μου απαντήσετε. Τώρα, η άλλη μου ερώτηση αφορά αυτό το σύστημα προειδοποίησης που έχουμε και στην ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Εάν κατάλαβα καλά, αυτό προβλέπεται μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος για τις υπηρεσίες των τομέα της δημόσιας δεν θα καλύπτονται. Γιατί ακριβώς αποκλείονται από την λογοδηγία. Αλλά όπως και ο πρόεδρο, έτσι και εγώ πιστεύω, ας αυτόν τον τομέα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα προειδοποίηση. Ε, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εάν παραδείγματο χάρη ένα γιατρό έχει χάσει την έγκριση άσκηση του επαγγέλματο σε ένα κράτος μέλος και θέλει να πάει σε ένα άλλο, δεν πρέπει να περάσει από αυτό το σύστημα. Πώ θα γίνεται, Έχετε εδώ κάτι κατά νου. Δεύτερη ερώτηση. είπατε ότι πρέπει να αναφέρετε για ποιες χώρες θα ισχύει αυτή η προεδοποίηση Και θα πρέπει να είμαστε κατά το περιοριστικοί όσον αφορά την επιλογή αυτών των κρατών. Αλλά όταν εγώ θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου γιατί βλέπω στη χώρα μου υπάρχει ε, κίνδυνος με, μία, με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ή κάτι. Εγώ δεν ξέρω πάντα. Σε ποια άλλη χώρα θέλουν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ήταν λογικότερο να υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνονται όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό να μην θεωρείτε ότι επιβαρύνει υπερβολικά το σύστημα. Παραδείγμα χάρη, ναι, έχω στη Γερμανία κάποιον θέλω να προειδοποιήσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Γιατί θα πρέπει να ειδοποιήσω μόνο τη Γαλλία και την Πολωνία αυτός μπορεί να πάει στο Λουξεμβούργο και στη Δανία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μου παρουσιάστηκε ακούγοντας την παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος η Χάντι Ρούιλε. Πολύ σύντομα. Ε, Όσον αφορά τη χρήση του συστήματος, ξέρω ότι στην αρχή στα διάφορα κράτη-μέλη υπήρχαν επιφυλάξεις. Δισταγμή αν θέλετε να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα όπως θα έπρεπε. Και αναρωτιέμαι τώρα, έχετε αριθμητικά στοιχεία πόσο χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη και δεύτερον τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και τι κάνετε εσείς ούτως ώστε να ε, μπορέσουν να μάθουν όλοι ότι μπορούν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Yeah. Um, Υπάρχει κάποιος άλλος. Θα ήθελα εσύ να απαντήσεις σε ερωτήσεις Μαρία. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσω με τη χρήση του συστήματος IMI πρώτα απ' όλα. Έχουμε 6.300 αρχές καταγεγραμμένες αυτή τη στιγμή στο σύστημα και αυξάνεται ο αριθμός τους. Μάλιστα πρόσφατα ε, συνδεθήκαμε και με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Το 10% όμως μόνο των αρχών αυτών πραγματικά ε, χρησιμοποιούν ενεργά το σύστημα. Είναι μεν ε, το 90% ε, γραμμένες, αλλά δεν το χρησιμοποιούν. Είτε γιατί δεν είχαν διασυνοριακές υποθέσεις, είτε γιατί δεν γνωρίζουν ακόμη τι πρέπει να κάνουμε το σύστημα. Οπότε πρώτα απ' όλα βλέπουμε γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα και δεύτερον προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα, Αριθμός αιτήσεων, αριθμός αιτημάτων που έχουμε λάβει ε, μέσω του IMI. Είναι γύρω στις 160 το μήνα που είναι και αυτό ε, μικρό ε, ποσοστό σε σχέση με τους τεράστιους τομείς υπηρεσιών και επαγγελματικών πρόσωπων που καλύπτονται. Κυρίω βλέπουμε δραστηριότητα σε επαγγελματικά προσόντα. Στι υπηρεσίε ε, σιγά σιγά βελτιώνονται τα πράγματα. Στην ετήσια έκθεση θα βρείτε περισσότερα αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια αντίγραφα στο τραπέζι εκεί μπροστά, αλλά και στην ιστοσελίδα του IMI μπορείτε να βρείτε πληροφορίε. Σε ό,τι αφορά τι προειδοποιήσει, το IMI μπορεί να κάνει σχεδόν οτιδήποτε έχει αποφασιστεί από πολιτική πλευρά ότι αποτελεί μια σωστή προσέγγιση. Δεν μπορούμε όμω εμεί να έχουμε ηγετικό ρόλο, ούτε να αφήσουμε την τεχνολογία να αποφασίζει τι θα πρέπει να γίνει. Πολύ σημαντικό βέβαια σε ένα τομέα όπω είναι οι προειδοποίησει, είναι το να υπάρχει μια στερή νομική βάση, γιατί μιλάμε για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορεί να αποφασίζει ότι α, ωραία καλή ιδέα είναι, ξεκινάμε. Πρέπει όλο αυτό να περιλαμβάνεται στην νομοθεσία και πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Με αυτή τη βάση λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το e-module, την ενότητα των προειδοποιήσεων σε οτιδήποτε άλλο ισχύ, σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς. Δεν έχουμε πρόβλημα τόσο με τα τεχνικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κάρτα, υπάρχουν ε, συζητήσεις αυτή τη στιγμή με τις επαγγελματικέ ενώσεις για να δούμε ποιο θα μπορούσε να είναι το καλύτερο μοντέλο μιας επαγγελματική κάρτας ε, ή επισκεπτηρίου και πώς θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό το σύστημα και το IMI. Εγώ νομίζω ότι είναι λογικό κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχουμε όλες αυτές τις αρχές που είναι καταχωρημένες στο σύστημά μας, έχουμε δηλαδή διάβλους επικοινωνίας. Όταν λοιπόν και εφόσον αποφασιστεί τι θα είναι ακριβώς αυτή η κάρτα, πώς θα λειτουργεί, φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί πάνω από έναν ενάμιση χρόνο για να προσαρμοστεί το σύστημα για αυτό το σκοπό επί του παρόντος έχουμε 35 επαγγέλματα. Αυτά τα 35 καλύπτονται στο σύστημα, αλλά έχουμε συμφωνήσει ήδη με τα κράτη-μέλη να διευρύνουμε το πεδίο ώστε να καλύψουμε και τα 800 ρυθμισμένα επαγγέλματα μέχρι τα τέλη του 2012. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο στόχο γιατί κάποια από αυτά τα 800 επαγγέλματα είναι ρυθμισμένα σε ένα ή δύο κράτη-μέλη μόνο. Άρα θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να ορίσει μια αρχή η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα των επαγγελμάτων που δεν είναι ρυθμισμένα στην χώρα τη συγκεκριμένη. Ίσως πάρει λίγο χρόνο αυτό. Τα περισσότερα όμω επαγγέλματα που χρειάζονται αυτό το σύστημα έχουν ήδη συμπεριληφθεί. Και μέχρι τα τέλη του 2010 θα μπορούμε να χειριστούμε όλα τα επαγγέλματα, όπω είπα. Μια τελευταία παρατήρηση για τι προειδοποιήσει. Η κυρία Γκέπχαρτ πολύ σωστά επισήμανε ότι οι υγειονομικέ υπηρεσίε δεν καλύπτονται από το σύστημα των προειδοποιήσεων. Όπω σα είπα, η προειδοποίηση πρέπει να βασίζεται σε μια νομική βάση, που είναι η οδηγία για τι υπηρεσίε. Εκεί δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίε υγεία. Τώρα, το θέμα κατά πόσον μια προειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται σε όλε τι χώρε ή μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμοχωρών. Ακούστε ή μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό χωρών. Ακούστε, προειδοποίηση για να σα δώσω ένα παράδειγμα έχει χρησιμοποιηθεί μία φορά μόνο πέρυσι συγκεκριμένα. Αφορούσε έναν ξεναγό ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα. Η χώρα, η συγκεκριμένη, γνώριζε ότι ο ξεναγός αυτό ε, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και σε δύο άλλες χώρες γι' αυτό αποφάσισε να στείλει προειδοποιήσει σε αυτές τις δύο χώρες μόνο. Εξαρτάται λοιπόν από την κατάσταση τελικά. Δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει αν ο ανασπάροχος υπηρεσίας θα παρέχει υπηρεσίες σε μία χώρα ή σε δύο ή σε όλες τις χώρες. Μία λύση είναι βέβαια να, ε, κάνεις, να τσεκάρει κανείς όλα τα τετραγωνίδια, αλλά μπορεί η υπηρεσία ή εν λόγω να αφορά ε, μία-δύο χώρες, οπότε η προειδοποίηση να είναι περιορισμένη. Αυτό ε, μια δυο χωρες οποτε η προεδοποιηση να ειναι περιορισμενη αυτο επιπλέον που προβλέπεται και στην οδηγία και τις υπηρεσίες, ώστε να λαμβάνεται πλήρως υπόψη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με το σύστημα αυτό τώρα μπορούμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, ό,τι έχει αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ακολουθούμε τις αποφάσεις εφόσον ληφθούν και τις τηρούμε. Ευχαριστώ. Uh, well, Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και που βέβαια ήρθατε και εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα σας προσκαλέσουμε σίγουρα ε, όταν θα έχει αναπτυχθεί το σύστημα και εξελιχθεί περισσότερο και επειδή συζητάμε και την αναγνώριση των προσόντων, η κυρία Βερνιό συγκεκριμένα με την ομάδα προβληματισμού ασχολείται πολύ ενεργά με αυτό το θέμα. Το ίδιο είχαμε κάνει άλλωστε και με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θυμάστε ότι τότε είχαμε συζητήσει και για τα εργαλεία εφαρμογής και διευκόλυνσης της ε, νομοθεσίας αυτής. Είναι λοιπόν πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό, γιατί αυτά τα εργαλεία πραγματικά θα βοηθήσουν πολύ στην ενιαία αγορά, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους, θα βοηθήσουν τους επαγγελματίε να μπορούν να μετακινούνται πιο ελεύθερα και να αντιμετωπίζουν κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την έλλειψη αποδοχής ε, προσόντων κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εσάς και τους συναδέλφους σας και ελπίζω να σας έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μας. Περιμένουμε τον Επίτροπο Ντάλι να έρθει, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί ε, φίλοι, οπότε σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης των συντονιστών. Θα ληφθούν, μάλλον ε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν θα σας διανεμηθούν όσοι ήθιστε. Προς ενημέρωσή σας να πω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν η Επιτροπή να αναλάβει την σύνταξη δύο γνωμοδοτήσεων μη νομοθετικού περιεχομένου. Πρώτη, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, εισηγητή από του Σοσιαλιστέ. Και δεύτερο, εμπόδια για τι επενδύσει και το εμπόριο, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, Διεθνής, ε, η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, εισηγητή από το ΕΛΚ πάντω. Και υπάρχουν κάποια άλλα θέματα για τα οποία δεν θα γνωμοδοτήσουμε. Θα δείτε ποια είναι αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι οι συντονιστέ μα αντιλαμβάνονται το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα εργασία που έχουμε στο μέλλον. Άρα θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία και να δώσουμε προτεραιότητα για τις βασικές ευθύνες και αρμόδια της Επιτροπής μας. Επιβεβαιώθηκε επίσης και χαίρομαι πολύ που θα είστε κυρία Σφέσον η συγγήτρια για τη στρατηγική για την καταναλωτική πολιτική, πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Επίσης αποφασίσαμε να υποβάλουμε ένα αίτημα για νέα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ως απάντηση στα Solvage Reports και στον ε, πίνακα επιδόσεων ε, το scoreboard που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά χωρίς πρόβλημα. Επίσης, αναμένουμε από την Κομισιόν μια πολύ σημαντική πρόταση για κάποιες οδηγίες. Κύριε για παραδείγματο χάρη που εργάζεται για τα εμπορεύματα, για τα αγαθά, νομίζω 9 οδηγίες θα συμπεριληφθούν. Και θα έχουμε για μια ξεχωριστή έκθεση Έχουμε διαπραγματεύσει και με άλλες επιτροπές. Ενημέρωσα τους συντονιστές ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων δέχτηκε την ενισχυμένη συνεργασία μαζί μας για τις εκθέσεις πεναλλακτική επίλυσης διαφορών. Επίσης, συζητούμε με την Οικονομική Επιτροπή τις τελικές διευθετήσεις για να έχουμε υποκλειστική αρμοδιότητα για τους τομείς της καταναλωτικής προστασίας ό,τι αφορά ε, τις ε, συμβάσεις ε, πίστοσης για τα ακίνητα, τα στεγαστικά δάνεια ουσιαστικά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο φόρουμ της ενιαίας αγοράς. 3 και 4 Οκτωβρίου στην Κρακοβία, με μεγάλη υποστήριξη από την Πολωνική Προεδρία. Θα είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εκδήλωση για πρώτη φορά μετά τη δρομολόγηση έκθεση για την ενιαία αγορά και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ε, κοινοβουλευτικέ αρχές ε, να επιτρέψουν να συμμετάσχει μια μεγάλη αντιπροσωπεία και από άλλες επιτροπές, αλλά να είναι μεγάλη η παρουσία της δικής μας επιτροπής. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες στο ημερολογιό σας και επίσης θα υπάρξει διακοινοβουλευτική συνάντηση με το Πολωνικό Κοινοβούλιο στις 10 και 11 Οκτωβρίου με εστίαση στα ζητήματα της ε, εσωτερικής αγοράς. Αυτή είναι η προτεραιότητά τους άλλωστε. Αυτές είναι οι κύριες ανακοινώσεις που ήθελα να κάνω. Και τέλος, κύριος Ρέπο ήρθε στους συντονιστές και μας μίλησε για τις τροποποίησεις του κανονισμού για την συνεργασία των καταναλωτών. Να καλώς όρισε τον Επίτροπο, που είναι και ένα από τα θέματα που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Χθες ε, ψηφίσαμε κύριος Ρέπου ζήτησε έγκριση από τους συντονιστές για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Συμφώνησαν οι συντονιστές, είναι έκτακτες οι συνθήκες σε σχέση με την πρόταση αυτή. Πρόκειται για μια σχετικά μικρή τροποποίηση και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε σύντομα να συμφωνήσουμε και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Μια καλή είδηση προς την Κομισιόν λοιπόν αυτή. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Έφτασε ο Τζον Ντάλι, τον χαιρετίζω για μια ακόμη φορά. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Ντάλι στην Επιτροπή μας. Θα μας μιλήσετε σήμερα για το πρόγραμμα εργασίας σας σε πολύ σημαντικό τομέα πολιτικής αυτών που είναι στην αρμοδιότητά του. Όλα τα μέλη φαντάζομαι έχετε τον πίνακα με τις πρωτοβουλίες του κύριου Ντάλι. κυρία Σβένσον, όπως είπα και πριν, είναι η συγγήτρια για την καταναλωτική στρατηγική έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Φαντάζομαι ότι η κυρία Σβένσον θα θέλει να θέσει ερωτήσει στον κύριο Ντάλι. Κύριε Ντάλι, σας δίνω λοιπόν ευχαρίστω τον λόγο για να μας μιλήσετε για τα σχέδιά σας. Ευχαριστώ πολύ και λυπούμε για την ολιγόλεπτη καθυστέρησή μου. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να συζητήσουμε τα σχετικά με τον τομέα μου μαζί σας. Πριν από κανένα χρόνο συναντηθήκαμε και από τότε γίνεται όλο και πιο σαφές ε, ότι η ε, Ευρώπη χρειάζεται νέες πηγές ανάπτυξης και επομένως ε, η καταναλωτική πολιτική είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να οθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τους στόχους του 2020. Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε την μεγάλη καταναλωτική δύναμη της Ευρώπης που συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ΑΕΠ γνωρίζουμε ότι μέσω της καταναλωτικής πολιτικής μπορούμε να οθήσουμε την ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν περισσότερο από ποτέ πιστεύω ότι ε, οι δυνατοί και καλά προστατευμένοι καταναλωτές μπορούν μόνο προστιθέμενη αξία να δώσουν στην ε, ενιαία αγορά. Πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως, η ενδυνάμωση δηλαδή πρώτα, είναι ε, ε, ένα σημαντικότατο στοιχείο. Είναι ακριβώς αυτό που βάζει τους καταναλωτές ε, στο κέντρο της εσωτερικής αγοράς και δεν αναφέρομαι εδώ μονάχα σε δικαιώματα των καταναλωτών. Αναφέρομαι στην ε, οικοδόμηση ενός γενικότερου περιβάλλοντος ε, μέσα στο οποίο θα αισθάνονται οι καταναλωτές άνετα. Σημαίνει ότι θα ε, έχουν από τη μία πλευρά οι καταναλωτές δυνατότητα πρόσβασης όχι μόνο σε καταναλωτικά αγαθά αλλά και σε οτιδήποτε άλλο προσφέρει η ενιαία αγορά. Σημαίνει επίσης ότι οι καταναλωτές θα βασίζονται στην αρχή ε, της ασφαλείας ε, και θα είναι σε θέση οποτεδήποτε δεν αισθάνονται ασφαλείς να ε, προσφεύγουν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο έτσι ώστε να λύνεται οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται. Αναφέρομαι επίσης σε μια οικοδόμηση αγοράς η οποία θα βασίζεται στην καινοτομία και ε, ότι οι φορείς της αγοράς θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα των καταναλωτών. Γι' αυτό ακριβώς ετοιμάζουμε μια νέα ε, στρατηγική για την καταναλωτική πολιτική και συζητιέται βέβαια στα πλαίσια του επερχόμενου προγράμματος. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος προσπαθούμε να εξεύρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις ε, έτσι ώστε το προσχέδιο τη στρατηγική στρατηγικής ε, για την καταναλωτική πολιτική να είναι ε, το καλύτερο δυνατό. Μαζί με την Επίτροπο ε, Ρέντινγκ συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να επιτύχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καταναλωτών. Θα ήθελα πέρα από την αναφορά σε παρούσες διεργασίες και πρωτοβουλίες να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αρχές και ιδέες και βεβαίως θα ήθελα και ανάδραση, θα ήθελα feedback από εσάς. Πρόσφατα σε ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρθηκε η ευαισθησία της απέναντι στα προβλήματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ο βασιλέας της ε, ε, εσωτερικής ε, αγοράς και όλοι οι καταναλωτές ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ε, να ενδυναμώσουν την παρουσία τους αλλά και τα δικαιώματά τους ε, στην εσωτερική ενιαία αυτή αγορά. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα για καλή πληροφόρηση, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, δυνατότητα επιστροφής προϊόντων, επίλυσης διαφορών κτλ. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους εύκολα κατανοήσιμη πληροφόρηση, αναλυτική πληροφόρηση επίσης, οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα σε μια ε, όλο ένα και πιο προκλητική ας πούμε και αναπτυσσόμενη αγορά ερχόμαστε σε επαφή και με τις ε, οργανώσεις των καταναλωτών, γιατί αυτή η σχέση είναι σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι η νέα μας στρατηγική θα στοχεύει και στην οικοδόμηση αλλά και την στήριξη ισχυρών καταναλωτικών οργανώσεων, οργανώσεων των καταναλωτών ε, που ε, παρουσιάζουν μέσω των θέσεών τους ενδιαφέρον και για τους καταναλωτές αλλά και για τους για όσους ε, δημιουργούν προγράμματα και λαμβάνουν αποφάσεις. Τέλος, ως ε, ε, υπεύθυνο για την καταναλωτική πολιτική σας βεβαιώ ότι θα συνεχίσω την ε, πολιτική βάση της οποίας ο καταναλωτής ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί στην ουσία όλες οι στρατηγικές, όλες οι κεντρικές στρατηγικές στοχεύουν τελικά στον καταναλωτή και στον πολίτη. Σας βεβαιώ επίσης ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην ενιαία εσωτερική αγορά θα γίνεται με κύριο γνώμονα και κύριο μέλημα των ε, πολίτη. Η έκθεση του καθηγητού κ. Μόντι ε, ε, αποτελεί βάση της εργασίας μας βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι και από αυτά που σας λέω και από αυτά που γνωρίζετε ότι η σπορά έχει γίνει και μάλιστα πολλαπλώς. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να μεγαλώσουν τα φυτά και βεβαίως να προχωρήσουμε στη συγκομιδή. Στις 16 Μαΐου ε, έγινε μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Κοινοβούλιο. Ε, κατεδείχθη ακριβώς η σημασία ε, της ε, προστασίας των καταναλωτών κυρίως όσον αφορά τις διασυνοριακές και τις επιγραμμικές συναλλαγές. Ε, υπεγραμμίστη η σημασία επίσης της μελλοντικής πρότασης για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ε, όλες αυτές ε, οι δυνατότητες ADR, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικές και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Όσον αφορά το θέμα αυτό, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε ότι έχουμε λάβει πάνω από 200 απαντήσεις από οργανώσεις οργανωμένους ε, ε, φορείς ε, που καταδεικνύει ακριβώς το ενδιαφέρον των καταναλωτών για θέματα αυτά. Επίσης, Σύντομα θα υπάρξει ένα πλαίσιο οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών αλλά επίσης και μια ειδική αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσον αφορά τώρα τις συλλογικές ε, προσφορές πρέπει να σας πω ότι οι απαντήσεις που είχαμε ήταν πάρα πολλές, ε, πολλές ε, χιλιάδες και επομένως μέχρι το τέλος του έτους σε συνεργασία με τον Επίτροπο Αλμούνια θα υποβάλουμε προτάσεις. Η προστασία όσον αφορά τα προϊόντα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς προχωρούμε στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των τροφίμων και βρισκόμαστε τώρα στην μελέτη μελέτη επιπτώσεων. Στοχεύω ε, μαζί με τον Επίτροπο Νταγιάννη ε, να υποβάλουμε στο δεύτερο εξάμεινο μία ανακοίνωση σχετικά με την ορθότερη επιτήρηση της αγοράς θεωρούμε ότι η αγορά αυτή θα πρέπει να είναι ε, προστατευτική για τους καταναλωτές, ε, να βοηθάει τις ε, επιχειρήσεις και επομένως να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Κατά αυτήν την έννοια θεωρώ ότι η έκθεση Αλντεμόζα είναι εξαιρετική εργασία και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή. Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη διεθνή συνεργασία κυρίως με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ε, και μάλιστα ε, στην επίσκεψη υψηλού επίπεδου ε, στην Κίνα κατά την οποία συμμετείχαμε στην υψηλού επίπεδου διμερή συνάντηση συζητήσαμε όλα τα θέματα. Αυτά. Όσον αφορά τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες πρέπει να σας πω ότι τα ECCs έχει, έχουν μπει σε τελική φάση. Σύμφωνα με το, με το ευρωμαρό, ευρωβαρόμετρο πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερος γνωστή σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και στην οποία πραγματικά εναποθέτουν πάρα πολλές ελπίδες. Ε, θεωρούμε ότι τα ίδια τα ECCs μπορούν να βοηθήσουν και μπορούμε περαιτέρω να οργανώσουμε τα δίκτυα αυτά έτσι ώστε πραγματικά να απαντήσουμε και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Η συνεργασία ε, των δικτύων ε, καταναλωτών ε, πραγματικά έχουν ενδυναμωθεί και ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο μέσα από την ενίσχυση και των εθνικών δομών που ήδη υπάρχουν και η προσπάθειά μας όσον αφορά την συμμόρφωση των προϊόντων έχει αρχίσει και καρποφορεί. Ε, ξεκινούμε επίσης και μία ανεξάρτητη, ε, ε, ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης της οδηγίας αυτής. Πάντως θεωρώ ότι χρειάζεται αντικειμενικά να αναλύσουμε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται και πού ακριβώς πρέπει να ενισχυθεί το πλαίσιο αυτό έτσι ώστε καλύτερα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών. Σαν Επίτροπος υπεύθυνο ε, για τους καταναλωτές και την καταναλωτική πολιτική, ε, έχω προσπαθήσει σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ε, που καλύπτονται από την εργασία των συναδέλφων μου του Κολεγίου των Επιτρόπων να ενσωματώσω την καταναλωτική πολιτική η εφαρμογή των ε, οδηγιών ε, οπωσδήποτε, ε, οπωσδήποτε εξαρτάται και από την δυνατότητα παροχής πόρων καθώς επίσης και από την διαφάνεια. Μαζί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να πω ότι η συνεργασία είναι πολύ καλή. Και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτή Ευρωπαϊκής είναι η οδηγία για τις ε, συμβάσεις ε, ε, ακινήτων, υποθηκών και δανείων. Το σημαντικό βέβαια όλων αυτών που έχω πει μέχρι τώρα είναι οι πράξεις μας τελικά να φτάνουν στους καταναλωτές, να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο. Όσον αφορά την ψηφιακή ατζέντα, εγώ πάντα ήμουν υπέρ της ε, ε, απόλυτης προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, των προσωπικών δεδομένων των πολιτών ε, και επομένως μιας διαδικασίας η οποία μόνο καλά θα τους προσφέρει ε, και δεν θα αφήνει περιθώρια για απατηλές συμπεριφορές, απάτες και γενικότερα δεν θα αφήνει περιθώρια ε, να εξαπατηθούν ε, οι καταναλωτές. Κατά αυτήν την έννοια περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία τα αποτελέσματα πολλών εργασιών και μελετών που έχουν ξεκινήσει ε, ε, σχετικά με τα θέματα αυτά. Ε, όσον αφορά τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce, ε, μας απασχολεί πάρα πολύ. Σε συνεργασία και με άλλους επιτρόπους ε, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν την δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου να έχουν καλύτερες υπηρεσίες και σε καλύτερες τιμές. Όσον αφορά τα, τις τηλεφωνικές υπηρεσίες επίσης προσπαθούμε να προωθήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε μόνο ωφέλη να προκύψουν για τους καταναλωτές καταναλωτές. Επίσης έχουμε ε, εισαγάγει την ε, ε, κατάσταση περιβαλλοντικής προστασίας όσον αφορά το λιανικό εμπόριο και θεωρούμε ότι αυτή είναι μια πολύ καλή διαδικασία πιστεύω ότι όλες, ε, ε, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει τροποποίηση των κανόνων θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ε, καταναλωτές έτσι ώστε να μην προκύπτουν ζημίες για τους καταναλωτές. Τέλος, σε συνεργασία με την κυρία Ρέντινγκ έχουμε προχωρήσει πολύ την εργασία μας όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις συμβάσεων και πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι βεβαίως να να ε, καταδείξουμε για μία ακόμα φορά πώς έχει ενσωματωθεί η καταναλωτική πολιτική σε όλες τις κεντρικές πολιτικές ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάρτιο δημοσιεύθηκε το πέμπτο scoreboard για τους καταναλωτές σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, η διάσκεψη η οποία οργανώθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο σαφώς κατέδειξε ότι ε, μέσω των νέων στρατηγικών ε, κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών έτσι ώστε ε, να ολοκληρώσουμε οι διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει και να οδηγηθούμε ορθότερα προς το μέλλον. Το σημαντικό είναι να καταρτήσουμε, και στρέφονται τώρα προς το μέλλον, να καταρτήσουμε λέγω το καλύτερο δυνατό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά να γνωρίζουν και πώς να τα χρησιμοποιήσουν και πώς να τα επιτύχουν. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν φτάσουμε στο σημείο αυτό, τότε δεν θα έχουμε επιτύχει στην καταναλωτική μας πολιτική. Η έρευνα για την ενδυνάμωση των καταναλωτών μας έχει δώσει πολύ σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την ε, κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πληροφόρησης των καταναλωτών επίσης μας έδωσε πανοπλία ε, ε, όπλων έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες ιδιαίτερες καταστάσεις που παρουσιάζονται στην αγορά. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο προϋπολογισμός για την καταναλωτική πολιτική θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί ίδιος και οπωσδήποτε να μην μειωθεί. Αγαπητοί φίλοι, Είμαι βέβαιος, ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει αλλάξει ούτε μία κεραία από αυτά που σας έλεγα όταν ξεκίνησα την ε, θητεία μου όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Επίσης ε, βασίζομαι στην καλή και δυνατή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή σας, στην οποία εξακολουθώ να βασίζομαι και θέλω να βασίζομαι και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Well, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε γιατί καλύψατε ένα ευρύτατο φάσμα στην παρουσίασή σας. Θέλουμε πάντοτε να σας ενθαρρύνουμε να είστε ένας πρωταθλητής υπέρ των καταναλωτών και αυτό δείχνει και η φιλόδοξη ατζέντα σας. Φυσικά και τη στηρίζουμε ένθερμα. Έχουμε και εμείς ε, κάποια σχέδια δικά μας για να συμπληρώσουμε το δικό σας έργο. Χαίρομαι επίσης που ανακοινώσετε ότι θα ξεκινήσετε να ε, χαράστηκε μία ε, στρατηγική για τους καταναλωτές, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά αυτή την έρευνα για την δυνάμωση των καταναλωτών, το empowerment ε, δεν νομίζω είχε παρουσιαστεί εκ των προτέρων σε εμά. Αυτό είναι πολύ καλό λοιπόν. Δεν ξέρω ποιες να θέλουν να ρωτήσουν τον Επίτροπο, αλλά να κάνω μια πρόταση. Νομίζω καλό θα ήταν οι εισηγητέ που εργάζονται για τα θέματα που αφορούν του καταναλωτέ. Εσεί αναφερθήκατε σε αρκετά θέματα που σχετίζονται με του καταναλωτέ. Θα ήταν ίσω καλό να είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το λόγο και να ακολουθήσουν άλλοι συνάδελφοι, αν συμφωνούν οι συντονιστέ. Νομίζω θα είναι έτσι μια καλή αλλαγή στι διαδικασίε μα. Οι συγητές λοιπόν και τον κύριο Αρία τον συμπεριλάβω για την ψηφιακή οικονομία γιατί αναφέρθηκε και αυτό το θέμα. Έχω λοιπόν την κυρία Σβένσον, πρώτη, Σαλντεμόζε επίσης, κύριος Ροσφόρ, κυρία Ράπτη. Α, θέλετε, ωραία. Εντάξει, και Αρίας. Είναι οι πρώτοι ομιλητές. Πέντε συγητέ, δηλαδή ξεκινούν και μετά ΣΦΑΠ, Γκέρχαρτ, Γκέπχαρτ και Κορέα Ντεκάμπος. Και όποιος άλλος θέλει να προσθέσει τον κατάλογο. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε όλους. Κυρία Σβένσο, πρώτη ερωτήσεις από πλευρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι προσβλέπουμε ανυπομονησία στη συνεργασία με τους συναδέλφους μας εδώ από την Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Ντάλι που ήρθε και μας μίλησε σήμερα εδώ και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για ένα πληρέστατο πρόγραμμα εργασίας που μας υποβάλλει. Όπως είπε και ο πρόεδρος, είμαι και εγώ πεπισμένη ότι έχουμε το ίδιο όραμα, την ίδια δέσμευση υπέρ των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχω κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα να θέσω στον Επίτροπο. Το Κοινοβούλιο σχεδιάζει να εκπονήσει έκθεση για μια στρατηγική για την καταναλωτική πολιτική. είχαμε και την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν μπορούμε, ε, ούτε και είναι και ευκταίο, να έχουμε μια πλήρη εναρμόνιση. Επίσης λάβαμε μια δημοσίευση από την Κομισιόν που κάνει λόγο για 12 βασικούς τομείς ε, πολιτικής για την ενιαία ε, Single Market Act, για την πράξη για την αγορά. Ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα, τι θα περιλάβετε στην προτινόμενη σα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών για το 2013 και μετά. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Εσωτερική αγορά. Νέα επικοινωνιακά εργαλεία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, μάλλον στους Ευρωπαίους καταναλωτές προσφέρονται όλο και νέα προϊόντα, όλο και νέες υπηρεσίες. Αλλά υπάρχουν και καταγγελίες και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ευοδοθούν καταγγελίες των καταναλωτών. Η ευρωπαϊκή οικονομία εξελίσσεται, προχωρά και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είμαι βέβαιη ότι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτή την προσέγγιση. Μέχρι στιγμής όμως το έργο της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ αφορούσε πιο πολύ τις διαδικασίες και όχι τόσο τον καθορισμό στόχων θα πρέπει να ενσωματώσουμε την διάσταση των καταναλωτών σε άλλες πτυχές. Την εκπαίδευση, δικαιώματα στην αγορά κτλ. Νομίζω ότι καλά είναι όλα αυτά που μας είπατε, αλλά χρειαζόμαστε πιο ισχυρά μέτρα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους αυτούς. Να βάλουμε τους καταναλωτές στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ τώρα Φεβρουαρίου και Απριλίου ε, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ οργάνωσε διαβουλεύσεις για κάποιες κοινέ νομικές αρχές σε ό,τι αφορά τις ε, συλλογικές προσφυγές. Και προσπάθησαμε να δούμε πώς θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί και στα νομικά συστήματα των 27 κρατών μελών. Σχεδιάζεται να λάβετε ειδικά συγκεκριμένα μέτρα. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις διαδικασίες διαβούλευσης. Και σε ό,τι αφορά το Single Market Act, διακόπτει ο πρόεδρος, ξέρετε πρέπει να ρωτήσουν και άλλοι, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να είστε λίγο πιο σύντομοι τις ερωτήσεις σας, αλλιώς δεν πρόκειται να προλάβουν οι συνάδελφοι να ρωτήσουν τα δικά τους ερωτήματα. Άλλωστε, όσοι εισηγήτρια θα έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε κάποια από αυτά τα θέματα και στη συνέχεια. Ναι, έχω ερωτήσει, λέει κυρία Σβένσον, έχω και άλλε ερωτήσει, αλλά φυσικά μπορώ να τι θέσω αργότερα ίσω ε, ή σε κάποια άλλη ευκαιρία. Είμαι βέβαια ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Θα ήθελα να ακούσω βέβαια και τι απόψει των συναδέλφων για να έχω την ευρύτατη δυνατή στήριξη για την έκθεση αυτή. Άρα σταματώ εδώ προς το παρόν. Θα μπορούσατε να τις ε, στείλετε στον κύριο Ντάλτσα ερωτήσεις σας. Κύριε Σαλντεμόζη, είναι επόμενη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντάλη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Δείχνεται πάρα πολύ δέσμευση για την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και αυτό με χαροποιεί. Εγώ εργάζομαι στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων και χαίρομαι που έχετε κατά νου να αναθεωρήσετε την Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Έχετε σκεφτεί πού θα ενταχθεί αυτή η αναθεώρηση δηλαδή θα αναθεωρηθεί ως έχει ή μέσα στα πλαίσια του νο, νέ, νέου νομοθετικού πλαισίου. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ε, εποπτείας στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς εκεί και τα κράτη-μέλη μας λένε ότι δεν έχουν τα χρήματα, τους λείπουν τα χρήματα Ε, εσείς έχετε σκεφτεί ως Κομισιόν πώς μπορεί να υπάρχουν περισσότερα χρήματα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων. Ευχαριστώ κύριε Ζωσφά. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Χάρηκα πάρα πολύ που έχετε αυτή τη φιλοδοξία και την ευκαιρία όπως ελέγχθη να ε, προωθήσετε την προστασία του καταναλωτή με τη λεγόμενη Single Market Act που θα υπάρξει φέτος. Είναι πολύ καλό που προσπαθείτε να έχετε μια γρήγορη οδηγία στον τομέα αυτών. Θα ήθελα σε ερώτηση το εσωτερικό αυτού του σχεδίου σας υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση που θα πρέπει να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Δηλαδή, να αναθεώρηση οδηγίας για τα πακέτα ταξιδιών. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλή εφαρμογή της ε, βούλησης, της αύξησης προστασίας των ε, καταναλωτών γιατί υπάρχουν πολλές ικανοποιήσεις και θα μπορούσε αυτό να ε, αναπτύξει την εσωτερική αγορά γιατί αυτή τη στιγμή η ελάχιστη εναρμόνιση οδηγεί σε πάρα πολύ υψηλό κόστος στις εταιρείες που θέλουν να προσαρμοστούν στην εσωτερική αγορά. Εκτός αυτού, η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής προβλέπεται για τα μέσα του 2011 και φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση θα την έχουμε αργότερα, θα ήθελα να ξέρω την δική σας άποψη και πώς συνεργάζεστε με τους αδέλφους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Νταλή για την παρουσία σας εδώ σήμερα και την εργασία που κάνετε μέχρι τώρα. Το θέμα μου είναι οι συλλογικές προσφυγές. Ένα θέμα που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει ανοιχτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην πατρίδα μου στην Ελλάδα λέμε μία παροιμία ότι όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει. Εδώ εσείς είστε τρεις επίτροποι που έχετε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Αυτό λιγάκι με ανησυχεί και με ανησυχεί διότι Χτες ήταν εδώ η συνάδελφό σας, η κυρία Ρέντινγκ, δεν είχα την ευκαιρία να τη ρωτήσω. Ε, αισθάνθηκα όμως ότι έχει μια πιο μακρινή απόσταση από τους καταναλωτές από ότι εσείς, έτσι όπως μας περιγράψατε τη θέση σας σήμερα εδώ. Και αυτό με ανησυχεί. Ε, νομίζω ότι τους καταναλωτές δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τους βλέπουμε με υποψία πρέπει να τους βλέπουμε θετικά. Ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον είστε διατεθειμένος να πιέσετε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, να πιέσετε τους συναδέλφους σας, ε, ώστε να έχουμε μια ανακοίνωση ως το τέλος του χρόνου, που όμως μέσα στην ανακοίνωση αυτή θα είναι σαφής η πρόθεση για νομοθετική πρωτοβουλία μέσα στο 12. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι μαζί μας, κυρίως ε, την παρουσία της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ στην ομάδα εργασίας για την Δροματική διοκτησία. Πολύ επικοδομητική συνεργασία μας. Δύο ερωτήσεις. Την πρώτη ε, την έκανε ο κύριος Ροσφόρ βέβαια σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο, που είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αν θέλουμε να ε, υπάρχει εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. <clears throat> Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο παραπάνω σε αυτό, κύριε Επίτροπε. Δεύτερον, σε μια από τι συνεδριάσει τη ομάδα εργασίας, είπαμε ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ έχει κάνει μια μελέτη για τι δυνατότητε του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι ίσως χάνουμε κάποιες ευκαιρίες στην Ευρώπη ε, που θα μπορούσαμε να έχουμε αποκομίσει μεγαλύτερα ωφέλη από αυτό το σύστημα. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο κι εσείς ε, πότε θα είναι έτοιμη αυτή η μελέτη και λίγο να επεκταθείτε πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ηγητές. Θα παρακαλώ στον κύριο Ντάλη να απαντήσει. Well, with regards ε, to the harmonization Όσον αφορά τα θέματα της εναρμόνισης ε, της νομοθεσίας, ξέρετε ποιες είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά. Αυτές οι δυσκολίες προέρχονται κυρίως από τις οργανώσεις καταναλωτές στις ε, ανεπτυγμένες χώρες που φοβούνται ότι η εναρμόνιση θα σημαίνει τελικά ενδεχομένως μείωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις χώρες τους δικαιώματα που κέρδισαν με τεράστιες προσπάθειες στην περασμένη δεκαετία. NGOs whenever Ήμουνα στη Ρουμανία πρόσφατα και συνάντησα ανθρώπους από τις, ε, από τις ε, οργανώσεις των καταναλωτών και μου λέγανε μα γιατί δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα όπως στη Σουηδία και τους είπα κοιτάξτε να δείτε αυτά τα δικαιώματα αποκτούνται με μάχες και με αγώνες μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα πρότυπα όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο ε, δικαιωμάτων χωρίς δηλαδή να εμπλακούμε σε θέματα εναρμόνισης που θα οδηγήσει σε έντονες ανησυχίες ίσως. Γιατί βέβαια υπάρχουν πολλά δικαιώματα που πρέπει να βελτιωθούν. Θα πρέπει να δούμε όμως και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε εκείνα τα δικαιώματα που πιστεύουμε ότι έχουν ένα αποδεκτό Επίπεδο. Δηλαδή θα πούμε ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο για τούτο ή το άλλο δικαίωμα στην Ευρώπη. Αυτό και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όλοι σε αυτό το επίπεδο. Ιδανικά, εγώ είμαι υπέρ της αναμόνης των δικαιωμάτων, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα ενδυναμώσει την ενιαία αγορά. Και πιστεύω ότι μια ισχυρή ενιαία αγορά είναι προς όφελος των καταναλωτών. Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά είναι τελικά πολύ προς όφελος του καταναλωτή. Αυτό είναι ο τελικός μας και κύριος στόχος μας. Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε νομίζω σταδιακά. Και γι' αυτό όταν πρέπει να ορίσουμε τις προτεραιότητες, νομίζω ότι στην ομιλία μου κασαζόρισα τις προτεραιότητες που έχω. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, που Ασχολούμεθα με αυτό και με τις τριμερείς ε, συμφωνίες που έχουμε με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα και πρόσφατα ήταν ο Υπουργός ε, ο Αρμόδος από την Κίνα εδώ. Συνεργαζόμαστε μαζί τους, ε, όπως σας είπα και το θέμα αυτό. Ανέμπλεξα και αυτή την ιδέα της ασφάλειας στην πηγή. Προωθώ αυτό το θέμα ότι θα πρέπει να εργαστούμε όσο σκληρότερο μπορούμε για να είμαστε σίγουροι ότι η ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει εκεί από όπου ξεκινάμε και όχι να πρέπει να οργανώνουμε και να δαπανούμε για να ελέγχουμε την ασφάλεια καθ' όλη τη ε, διάρκεια της αλυσίδας. Εδώ δεν θέλω ότι δεν πρέπει να γίνεται τόπιν κανένα έλεγχο, αλλά η αρχική μα επένδυση θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική εάν τονίσουμε το θέμα τη ασφάλεια στην πηγή. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος που να σας πω ότι η ίδια η Κίνα ε, θέλει τώρα να προωθήσει την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει. Είναι λογικό αυτό. Γιατί και ήδη οι Κινέζοι αξίζουν ποιότητα όσο και εμείς. Εκτός αυτού, οικονομικά έχει απόλυτο νόημα κάτι τέτοιο. Μετά είναι το θέμα των προσφυγών. Ξέρετε ότι πιέζω για το θέμα αυτό. Εκτός από το θέμα της πρωτοβουλίας της συλλογικής προσφυγής, που προωθούμε με τον Επρό Δαλμούνια και Ρέντινγκ ε, έχουμε ξεκινήσει και ε, μία πρωτοβουλία για το ADR γιατί πιστεύω ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον παρατονική ε, καταναλωτή. Αυτό το θέμα των μικρών απαιτήσεων ε, είναι κάτι που πραγματικά αφορά πολλούς και έντονα και θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το τονέα και από κοινού νομίζω ότι θα μπορούμε να αποδώσουμε Μερικοί λένε ε, ότι γιατί εμείς αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούμε για τις επιχειρήσεις, για τους τομείς Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εγώ θέλω να συμφωνήσω αυτή την εναλλεκτική ε, δυνατότητα στους καταναλωτές. Να συγκεντρώσουμε λέει, την προσοχή μας στους καταναλωτές. Εάν ε, λειτουργήσει καλά, ας το αντιγράψουν κι άλλοι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα της ADR θα πρέπει να το παρουσιάσουμε καταρχήν στους καταναλωτές. Αλλιώς θα χάσουμε την ορμή που μπορούμε να έχουμε και θα αναβάλουμε χρόνια, για χρόνια την εφαρμογή οποιασδήποτε πρότασης μπορεί να γίνει σχετικά. Αυτή είναι η θέση μου και θα ήθελα να με βοηθήσετε, αν συμφωνείτε βέβαια. Επικοινωνία. Σημαντικότατο και πιστεύω ότι να αλλάξουμε τις στάσεις, να αλλάξουμε τις απόψεις είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ. Εργαζόμαστε πολύ. Εδώ και ενάμιση χρόνο που είμαι εδώ, πολλά έμαθα. Και βλέπω ότι θα πρέπει πραγματικά το κοινοβούλιο, βλέπω ότι προωθεί την νομοθεσία, τους κανονισμούς, αλλά όπως σας είπα και εισαγωγικά, όλα αυτά δεν θα έχουν κανένα νόημα αν δεν είναι μαζί μας οι καταναλωτές. Εάν δεν ξέρουν τι υπάρχει, εάν δεν ξέρουν πώς να εφαρμόσουν τα εργαλεία που τους δίνουμε στην προσωπική του ζωή, στην προσωπική τους υπόθεση, τους χάνουμε. Και αυτές είναι οι πληροφορίες που θέλουμε να βάσουμε στους αυτό είναι το πιο δύσκολο τμήμα της εργασίας μου. Γιατί έχω μακρά εμπειρία στην πολιτική και βλέπω ότι το να περάσει το μήνυμα απαιτεί συνεχή επανάληψη του μηνύματος. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια ανακοίνωση δεν αρκεί. Κάθε δύο μέρες πρέπει να το λέμε και το ξαναλέμε, το ξανά ξαναλέμε για εβδομάδες, για μήνες, ούτως ώστε να το ενστενιστούν. Όσον αφορά τα άλλα ερωτήματα της κυρίας Φένσον, Ευχαριστώ να έχουμε και μια κατηδία συνάντηση για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα γιατί χαιρετίζω οποιοδήποτε feedback μπορούμε να έχουμε. Όσον αφορά την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων που έθιξε η κυρία Σάλτερ Ομολογώ ότι η εμπειρία που είχαμε από την θεωρηθεί και παρόλο που είναι δυνατό να έρθει ε, και να συνενωθούν οι διάφορες ε, ε, διαδικασίες επιβολής της ασφάλειας, ότι αυτό ακριβώς λέω είναι ο στόχος μας. Ας είμαστε σίγουροι ότι όσον αφορά θέματα ασφαλείας, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Για να μην έχουμε κάποια προϊόνα που δεν πάνε ούτε εδώ ούτε εκεί και εξαφανίζονται. Είναι δύσκολο βέβαια να εξετάσει κανένα μεμονωμένα κάποια θέματα, γιατί ξεκινώντα από το ένα θέμα, περνάει στο άλλο, περνάει στο άλλο. και η οδηγία αυτή έχει ένα σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία αναζωογόνησης της ε, ε, νέας αγοράς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους πόρους κατά το δυνατόν βέλτιστα. Τι γίνεται με τα χρήματα. Εγώ στη Μάλτα ήμουν υπουργός οικονομικών 10 χρόνια. Ξέρω λοιπόν τη σημασία των χρημάτων. Ξέρουμε τους περιορισμούς που έχουμε για, στους προπολογισμούς μας. Και τώρα το εξετάζουμε και μέσα στα πλαίσια του νέου ε, χρηματοδοτικού πλαισίου. Καμιά φορά όταν συζητάμε για προπολογισμού σε αυτό το τομέα σε σχέση με προπολογισμού άλλων τομέων, εμείς μιλάμε για λίγα χρήματα. και παραβλέπετε το θέμα γι' αυτό πολλές φορές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι και να κάνουμε αφορά ανθρώπους και για να δαπανίσουμε χρήματα για να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση, είναι ικανοί και μάλιστα εμένα μου αρέσει ο όρος empowerment στα, στα αγγλικά, ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Αυτή η δυνατότητα που δίνουμε στον καταναλωτή είναι αυτό που κινεί την πολιτική μας. Εάν ο καταναλωτής δεν αγοράσει, δεν αντιδράσει μέσα στην αγορά, τι κάνουμε. Θα δαπανούσαμε χρήματα και πόρους άδικα. Λέω πάντως συναδέλφους και προσπαθώ να το επαναλάβω ότι στην πραγματικότητα εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονται στην αγορά κάθε ώρα. Αν όλοι αυτοί θα μπορούσαν να συνενωθούν, καταλαβαίνετε ποια θα ήταν η ισχύς της αγοράς των καταναλωτών. Πόσες πληροφορίες θα μπορέσουν έτσι να προωθηθούν προς τις εταιρείες που θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να ταιριάζουν στους καταναλωτέ. Και να έχουμε και εμείς αυτές τις πληροφορίες για να καταλαβαίνουμε καλύτερα ως νομοθέτες περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, όσον αφορά τις πληροφορίες, να προσπαθήσουμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και κάποια χρήματα, να βρούμε κάποια χρήματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κυρίως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα συστήματα είναι αποτελεσματικά. Γιατί το να μπορεί κανένας να κάνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα δεν είναι κοινοτυπία, είναι σημαντικό. Βεβαίως υπάρχουν ε, καθυστερήσεις και λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, όσον αφορά τα, πακέτα των ταξιδι... τα ταξιδιωτικά πακέτα, προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Βεβαίω, ένα από τα κεντρικότερα προβλήματα που έχουμε και που αντιμετωπίσα είναι ότι δεν είχαμε αρκετά αξιόπιστα στοιχεία για να κάνουμε τι ε, απαραίτητε αξιολογήσει όσον αφορά τι επιλογέ στρατηγική που είχαμε. Επίσης, ο Επίτροπος Κάλλας πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης όσον αφορά ε, την προστασία των ταξιδιωτών που έχουν πάρει απλά εισιτήρια και πακέτα ε, σε περίπτωση πτώχευσης ε, του ταξιδιωτικού γραφείου. Ξεκινήσαμε νομίζοντας ότι ήταν απλό το θέμα, αλλά τελικά καταλήξαμε σε δύσκολα εδάφη. Ελπίζω ότι θα τελειώσει το ζήτημα σύντομα όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή νομίζω ότι ήδη έχω ε, ε, δείξει ε, προς τα που κλείνω. Εγώ αναφέρθηκα σε ένα καθαρά ευρωπαϊκό πλαίσιο ευρωπαϊκής, συγγνώμη, ευρωπαϊκό πλαίσιο συλλογικής προσφυγής που θα διασφαλίζει την σωστή προοπτική, την συνεκτική γραμμή που θέλουμε να έχουμε, όπως είπα στη διαβούλευση Είχαμε πάρα πολλές απαντήσεις, πάρα πολλές απαντήσεις, 18.000. Ε, και πρέπει να σας πω ότι 6.000 είχαμε πάρει για την πρωτοβουλία για τον καπνό, δεν ξέρω τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Πάντως είχαμε μεγάλη ανταπόκριση και πρόκειται μια, για μια διεργασία την οποία πρέπει να προπεράσουμε, θα πρέπει να αναλύσουμε ε, όλα τα στοιχεία αυτά. Αλλά επ' αυτού δεν μπορώ να δεσμευτώ σε ημερομηνίες. Μέχρι το τέλος του χρόνου μπορώ να σας πω όμως ότι θα υπάρχει μια ανακοίνωση, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας. Στοχεύουμε να κινηθούμε γρήγορα και πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό αυτή την ανακοίνωση δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους. Ε, πάντως αρκεί να σας πω ότι και εγώ ο ίδιος αλλά και οι υπηρεσίες μου πραγματικά θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, και που, που πρέπει να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, και σε σχέση και με την ε, ADR, σε σχέση με την εναλλακτική επίλυση ε, διαφορών, ε, πρέπει να πω ότι εμείς προωθούμεθα προς, την, προς τη δυνατότητα προσφυγής και για επιγραμμικές υπηρεσίες, για online Θέλουμε να είμαστε proactive όσον αφορά τις διαδικασίες ε, συλλογικών ε, προσφυγών αλλά και ε, εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Το καλό είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια ευρυτάτη συζήτηση σχετικά με το προς τα που οδεύει το ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί εντάξει ο καθένας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ε, ε, θα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα βεβαίως να εκφράζεται ελεύθερα, αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τον οποιονδήποτε να λέει οτιδήποτε για οποιονδήποτε. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα είδος λογοδοσίας και θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ελέγχου. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμια. Συγγνώμη που μακρηγορώ. Μου λένε εδώ ότι η μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce ε, θα δημοσιοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε πολύ σύντομα να στριμώξουμε έναν ακόμα μικρό γύρο ερωτήσεων. Σίγουρα οι απαντήσεις σας κύριε Επίτροπε ήταν πληρέστατες. Θα βοηθήσει αυτό πολύ τους συγκητέ. Ε, έχω τη δυνατότητα να δώσω το λόγο ε, πάντω σε κάποιους ακόμη συναδέλφους, τους οποίους σας είχα αναγνώσει προηγουμένως. Ξεκινάμε λοιπόν τον κύριο Σφαμπ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, καλό είναι που παίρνω το λόγο στο δεύτερο γύρο Έχοντα ακούσει την απάντησή σας. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Αλλά πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ξεκάθαρες εξαγγελίε που κάνατε ενώπιον τη επιτροπή μα. Και απαντήσατε και σε ερωτήματα που δεν σας ετέθησαν. παραδείγματο χάρη το σύστημα B2B, ε, business to business, είπατε ότι υπάρχει μια εναλλακτική ε, λύση και σας ευχαριστώ που απαντήσατε. Φαντάζομαι ότι με τη δική σας ε, παρουσία όλα αυτά τα θέματα θα τα προασπίσετε στι Βρυξέλλες. Είναι αναζωογονητικό να σας ακούει κανεί να μιλάτε. Ένα άλλο θέμα, πνευματική διοκτησία. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο αλλά και η Κομισιόν έχουν προτείνει μια πολύ σημαντική στρατηγική. Νομίζω ότι η πνευματική ιδιοκτησία διαδραματίζει έναν σημαντικότατο ρόλο στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο και νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πνευματική ιδιοκτησία σε όλη τη νομοθεσία. Όταν λοιπόν υποβάλλεται κάποια πρόταση, ε, παραδείγματο χάρη για τη διαφήμιση σε σχέση με το τσιγάρο, θα έπρεπε και εκεί να λαμβάνονται υπόψη η διάσταση της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, ό,τι αφορά τώρα τα εμπορικά σήματα, την αντικατάσταση. Ε, η κυρία Ράπτη επίσης εξέφρασε την ανησυχία της πολλοί σκέφτονται τις συλλογικέ προσφυγές, αλλά εδώ μιλάμε για εναλλακτική επίλυση διαφορών, ADR, μιλάμε για μικρά ποσά. Είμαι πεπισμένος ότι η συλλογική προσφυγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση. Ο καταναλωτής δεν θέλει να έχει ένα πολύπλοκο εργαλείο, το αντίθετο θέλει. Υπάρχουν πάντως ε, εμπειρίες από διάφορα κράτη-μέλη. Είναι θετική η προσέγγισή σας και θα σας παρακαλούσα να κάνετε περισσότερα πράγματα στι Βρυξέλλες εδώ. Πρέπει να κάνουμε πράγματα για τους καταναλωτές. Μπορούμε να δράσουμε με ταχύ ρυθμούς και να καταλήξουμε σε κοινή θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι μπορούμε να στηριζόμαστε σε εσά. Κυρία Γκέπχαρτα. Πάντοτε είναι ωραίο να έπομε του κυρίου Σφάμπ γιατί τα λέει πρώτα αυτός και εγώ μετά έχω πιο εύκολη δουλειά. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πολύ που είστε δεσμευμένος υπέρ των δικαιωμάτων των καταναλωτών και συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι καλό είναι να υπάρχει εναλλακτική επίλυση διαφορών. Δεν είναι γραφειοκρατική ως διαδικασία, άρα μπορεί να είναι ταχεία και αποτελεσματική. Ταυτόχρονα όμως, Χρειαζόμαστε τη συλλογική προσφυγή, χρειαζόμαστε και τη συλλογική προσφυγή. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα με την ADR, την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Έλπιζα να μας πείτε ότι και αυτό το θέμα θα το ε, προχωρήσετε. Θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τυχημένα συστήματα. Μες στην Πορτογαλία, κοιτάζω τον κύριο Κορέα, τον συνάδελφο και στη Γερμανία έχουμε συστήματα για άλλους τομείς. Γιατί να μην μπορεί το ίδιο σύστημα να ισχύσει για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχω και ένα ερώτημα. Η κυρία Στανάλογα που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, αλλά ήθελε να θέσει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Με βάση μία μελέτη από μία Σλοβακική Ένωση Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, κατάλογης συστατικών από την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και το τι κανόνες ε, εφαρμόζονται για αυτά τα ε, συστατικά, για αυτόν τον κατάλογο των συστατικών. Δεν είναι ακριβώς στην αρμοδιότητά μας, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα με το κατά πόσον τα πρότυπα είναι ίδια με τα δικά μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ να αντιμετωπίσετε και αυτό το θέμα, όταν παραδείγματο χάρη οι προϋποθέσεις ή οι όροι ποιότητα είναι χαμηλότεροι και όταν δεν υπάρχει επαρκής προστασία των καταναλωτών σε αυτές τις χώρες. Ε, είπατε κάτι για τη Ρουμανία. Ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε περιπτώσεις ε, διάκρισης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και δεν θα πρέπει να έχουμε και πολίτες πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Οι συστάσεις, η σύνθεση των πρώτων πρέπει να είναι ίδια παντού κύριος Κορέια θέλει γρήγορα το λόγο. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Επιτροπός είναι υπέρ της ανάπτυξης αυτού του συστήματος ε, συλλογικών προσφυγών. Βέβαια καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να χωνέψετε, να επεξεργαστείτε το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Μετά από τις διαβουλεύσεις θα χρειαστείτε, λέτε, μέχρι το τέλος του χρόνου ε, μία περίοδο μέχρι ότου δημοσιεύσει την ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη ίσως να μην συμφωνούν πάντοτε με τις προθέσεις ε, της Ευρώπης των εθνών. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να περιμένει και ε, αισιόδοξο να περιμένουν να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Πρέπει να δείξετε μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Ω Επιτροπή πρέπει να παρενεβαίνετε περισσότερο. Δεν θα πρέπει να περιμένετε και να ελπίζετε ότι κάποιοι θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι α, ε, σύντομος όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να σας πω ότι απασχολεί πάρα πολύ τον Επιτρόπο Μπαρνιέ. Δουλεύει πολύ σκληρά για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουμε την καινοτομία μας, την ε, ε, πνευματική μας παραγωγή, την, ε, τις ευρεσιτεχνίες μας, τα πάντα. Απ' την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα τα οποία να είναι λογικά και να στέκουν και που τελικά θα διευκολύνουν την διεμπόρευση αυτών των ε, προϊόντων που θα βοηθήσουν τα προϊόντα να φτάσουν τελικά στους καταναλωτές. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τους ε, σωστούς κανόνες και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει το θέμα αυτό ενδελεχώς ε, στο εγγύ μέλλον. Όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή, είπα ότι συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ. βεβαίω χρειαζόμαστε δυνατότητα συλλογική προσφυγής, ε, γιατί αισθανόμαστε ότι είναι πραγματικά ε, κάτι πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι και συμπληρωματικό εργαλείο προς την εναλλακτική επίλυση διαφορών γιατί η ADR, η εναλλακτική επίλυση διαφορών από μόνη της ε, δεν στέκει ε, πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί με κάθε δυνατότητα επίλυσης διαφορών από την αρχή της διαδικασίας μέχρι το τέλος. Γι' αυτό ακριβώς ε, κινούμαστε και ε, ε, για τα δύο θέματα. Και λέω και εδώ ότι ναι, θέλουμε να προωθήσουμε την εναλλακτική επίλυση διαφορών, αλλά οπωσδήποτε και σε συνδυασμό με την δυνατότητα συλλογικής προσφυγής. Γιατί διαφορετικά δεν θα έχει πολύ μεγάλη έννοια. Τώρα, ε, διαφορά στη σύνθεση των προϊόντων και των προϊόντων εν γέννη μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής ε, Ευρώπης. Ναι, έχουμε διαπιστώσει μερικέ φορέ κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα διασφαλιστούν τα ελάχιστα πρότυπα. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και είναι αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει άμεσα και το ελέγχει. Η διατήρηση λοιπόν ελαχίστων προτύπων, minimum standards. Ε, και ακριβώς αυτό σας έλεγα προηγουμένως, ότι στη Ρουμανία ήρθα σε επαφή με οργανώσεις καταναλωτών ε, που ακριβώς ε, μου υπέβαλαν τέτοιου είδους αιτήματα, αναφέρθηκαν και σε προϊόντα, σε σύνθεση προϊόντων, και ε, επίσης αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο πολλές φορές στα ίδια πακέτα να περιλαμβάνονται διαφορετικά προϊόντα και αυτό είναι απατηλό ε, και μπορεί να οδηγήσει τους ε, καταναλωτές σε σφάλμα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που και μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ελαχίστων προτύπων. Uh, uh, όσον αφορά ε, την ε, προενεργητικότητα, την proactivity ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, ειδικά όσον αφορά το τομέα των προσφυγών, που είναι πραγματικά ένα τομέα στον οποίο επικεντρώνουμε τη σκέψη μας φέτος, ναι, νομίζω ότι είμαστε proactive και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καλές λύσεις και όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή και όσον αφορά την ίδια την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, που ήρθατε ε, σε εμά σήμερα το πρωί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Μας μιλήσατε για τη δουλειά σας και καταλαβαίνουμε βεβαίω ότι και εσεί δουλεύετε σκληρά, αλλά πρέπει να σα πω και να σα διαβεβαιώσω ότι και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως είναι οι συλλογικές προσφυγές, όπως είναι ε, η εναλλακτική επίλυση προσφορών. Έχουμε εισηγητές, έχουμε σκιώδεις εισηγητές, μιλάμε και δουλεύουμε για το πακέτο ταξιδιών και ε, ε, πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολλά και εμείς. Βλέπω βέβαια εδώ και πολλούς, ε, πολλές γνώριμες φυσιογνωμίες, ε, ε, ανθρώπους που τους βλέπουμε συχνά στη διάρκεια των εργασιών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Uh, so, um, και κύριοι, περνάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό πεδίο που έχει να κάνει με τους καταναλωτές και με την κοινωνία των πολιτών και με την τεχνολογία των πληροφοριών. Ε, σε πολύ λίγο, σε κανένα τέταρτο περίπου, θα έρθει η Επίτροπος Λικρούς. Μπορεί και να αργήσει, αλλά πιστεύω θα είναι εδώ. Βέβαια, ίσω να την ενδιαφέρει, έτσι πιστεύω, και το θέμα που θα συζητήσουμε. Α, στι 11.30 θα έρθει. Α, πολύ ωραία, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει λοιπόν η Επίτροπο Νέλη Κρού στις 11.30 θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είχαν αποφασίσει οι συντονιστέ ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον των εργασιών τη Επιτροπή μα και συγκεκριμένα ανατέθηκε η διεξαγωγή μια μελέτη με θέμα την ουδετερότητα του δικτύου. Είχαμε την προηγούμενη φορά ε, και τα δικαιώματα ε, των χρηστών. Είχαμε εκπονήσει και σχετική έκθεση στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. οποίο εργάζεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει να ξέρει διάφορες ε, εκφράσεις και είναι πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιήσει και να ξεμπερδέψει κανείς τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θελήσαμε κι εμείς να έχουμε αυτή τη μελέτη. Και έχουμε, ε, είπα, θέμα, είναι η ουδετερότητα του δικτύου, προκλήσεις και απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Θα ακούσουμε τη σχετική παρουσίαση. Να πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ θυμόμαι ότι εργαζόμουν ε, για κάποιον που μου έλεγε συνέχεια. Πού είναι το γλωσσάριό σου, πού είναι, πού είναι η ορολογία σου. Υπάρχουν όλα αυτά τα, τα αρχικά, οι συντομογραφίες. Θα σας τα πει όλα αυτά τα αρχικά ο μιλητής μας. Ε, ε, φαντάζομαι ότι κάποια θα μπορέσετε να τα αναγνωρίσετε, μπορείτε να κάνετε έτσι και ένα τεστ. Αλλά πιστεύω ότι η παρουσίασή του, όπως και η έκθεση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η ομάδα που συνέλα, συνέταξε την έκθεση είναι πάρα πολύ ειδική σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο Σκοτ Μάρκ είναι διευθυντής του WIC Consult που έχει έδρα τη Βόνη, θα μας μιλήσει για τη μελέτη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμπορ. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και έχω τη δυνατότητα να σας ε, μιλήσω αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Περάσουμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό το οποίο θα σας ε, περιγράψω σήμερα μετά από μια σύντομη εισαγωγή είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο και το οικονομικό υπόβαθρο περί ουδετερότητας δικτύου. Θα σας μιλήσω για τη διαφοροποίηση, την ποιοτική, δηλαδή και πώς, πώς μπορεί αυτό να σχετίζεται με τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει στην Επιτροπή σας. Και επίσης θα εστιάσω στις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, όχι σε ό,τι αφορά τη δομή της αγοράς μόνο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται και στις δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, ε, α, και μετά θα ολοκληρώσω με κάποιε στάσει. Είναι της αγωγή, να σα πω πρώτα απ' όλα ότι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα με την οποία εργαστήκαμε. Τζόναθαν Cave, Πίτερ Νόρν, μεταξύ αυτών. Εγώ προσωπικά έχω προσεγγίσει το ζήτημα από πολλές διαφορετικές σκοπιές ήμουν ε, αρμόδιος για θέματα τεχνολογίας ε, στο GTE που ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό τους ε, γραφείο στον τομέα των τεχνολογιών. Ασχολήθηκα με την τεχνολογική πολιτική στο FCC, εκεί συνάντησα και τον κύριο Χάρμπορ για πρώτη φορά και ήμουν και διευθυντής για μια συμφωνία ρυθμιστικών τεχνολογιών, regulatory, μάλλον οικονομιών, regulatory economy. Όπως λέω λοιπόν, είναι πολλές επιτυχίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και αφού τα είπα όλα αυτά, ας πάω στο επόμενο slide. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε τα εξής. Πώς ορίζουμε την ουδετερότητα Δεύτερον, τι ανησυχίε προκύπτουν. Και τρίτον, τι γνωστές, ε, τι, προβλήματα είναι γνωστά σήμερα. Για ορισμούς, πολλούς ε, μπορούμε να αναφέρουμε, πολλοί εφαρμόζονται. Ένα ορισμό είναι η ικανότητα και η δυνατότητα όλων των χρηστών του διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τη εφαρμογή επιλογή του. Μια άλλη ε, είναι ότι όλες οι κυκλοφορίες, όλη η κυκλοφορία στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα ανεξαρτήτως περιεχομένου ε, πηγής ή προορισμού. Τρίτος ορισμός, απουσία ε, μη εύλογης διάκρισης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ποιοτική διαφοροποίηση που είναι και στο επίκεντρο της συζήτησης για την ιδιαιτερότητα του δικτύου από μόνη της έχει και θετικές και αρνητικέ πτυχέ. Η ποιοτική διαφοροποίηση μπορεί να είναι θετική και να βοηθήσει και του καταναλωτέ και του παραγωγού ε, και χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο εδώ και καιρό. Επόμενη διαφάνεια. Οι παραβάσει του δικτύου. Υπάρχουν διάφοροι φόβοι. Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ε, επιρροή στο πεδίο ανταγωνισμού, Απειλέ κατά τη καινοτομία ή κατά της ελευθερίας έκφρασης ή κατά της συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Γνωρίζουν, καταλαβαίνουν οι καταναλωτές την υπηρεσία που τους προσφέρεται ή θέματα προσωπική ιδιωτικής σφαίρας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ανησυχίες που, αναφέρονται. Τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί κάποιε φορέ και των δύο πλευρών τα παρουσιάζουν ε, πολύ έτσι ε, μονόπλευρα, άσπρο ή μαύρο. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί αν λάβουμε ε, τα μη ε, κατάλληλα μέτρα θα κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τελικά ποιε είναι οι γνωστέ ε, βλάβε και σημείε που έχουμε εντοπίσει στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε μια δημόσια διαβούλευση με πολλές απαντήσεις. και ε, συγκεκριμένα από την ΜΠΕΡΕΚ, τον φορέα των τηλεπικοινωνιών. Και είδε ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ χρηστών του διαδικτύου, παροχών υπηρεσιών διαδικτύου και κατασκευαστών υποδομής που λέει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ε, με το άνοιγμα του διαδικτύου και την ουδετερότητα του δικτύου, ότι δεν βλέπουμε να υπάρχουν ενδείξεις να δείχνουν ότι υπάρχει ε, άδικη διάκριση και αυτό να βλάπτει καταναλωτές ή τον ανταγωνισμό και λένε ότι αυτή η γενική άποψη υποστηρίζεται από ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πόρισμα. Αν διαβάσετε τι απαντήσει και αν ρωτήσετε κόσμο, νομίζω ότι αυτό που σας ανάγνωσα συνοψίζει ποιε είναι οι απόψει των παρόχων. Υπήρξαν βέβαια καταγγελίες, κάποιες από αυτές ήταν αξιόπιστες σε σχέση με τους ε, φορείς κινητών υπηρεσιών που είτε μπλοκάριζαν είτε χρέωναν υπερβολικά το VoIP, τις φωνητικές ε, υπηρεσίες μέσω πρωτοκόλ. Ή επίσης μπλοκάριζαν ε, την ε, κυκλοφορία, παραδείγματος χάρη το file sharing. Είπαν όμως ότι αυτό μπορεί να μην αποτελεί παράβαση της ιδιαιτερότητας του διαδικτύου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές βέβαια προέβησαν σε κάποιες έρευνες. Ε, ε, το θέμα είναι τι θέλουμε τελικά. Λίγα είναι τα τεκμηριωμένα προβληματικά τέτοια κρούσματα στην Ευρώπη. Δεν φαίνεται να υπάρχει, να έχει καταδειχθεί ότι υπάρχει ένα σταθερό πρότυπο συστηματικής και καταχρηστικής διάκρισης, αλλά υπάρχουν ανησυχίες και νομίζω ότι πρέπει να ε, τις λάβουμε υπόψη γιατί είναι ανοιχτό τα ζητήματα για το μέλλον. Δηλαδή θα πρέπει να τα παραβλέψουμε. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα προβλήματα, αυτές τις ανησυχίες. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο τεχνολογικό υπόβαθρο θα καλύψω τη σουίτα πρωτοκόλλου διαδικτύου και τι αυτό σημαίνει ποιότητα υπηρεσία εμπειρία στο διαδίκτυο. Θα θυμάστε ότι για την ιδιαιτερότητα του δικτύου πολλοί ορισμοί έχουν να κάνουν με το αν ευνοείται κάποια κυκλοφορία σε βάρος κάποιας άλλης κυκλοφορίας. Και τι θα πει αυτό. Το διαδίκτυο, όπως βλέπετε εδώ, είναι μια διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική δικτύου όπως λέγεται, δηλαδή αποτελείται από στρώματα. Έχουμε τα κατώτερα στρώματα που βλέπουμε στο διάγραμμα που είναι πιο κοντά ε, στο φυσικό μέσο μεταφοράς και μετά τα ανώτερα στρώματα που είναι εφαρμογέ. Ο web browser δηλαδή που έχετε στον υπολογιστή σας για παράδειγμα είναι εφαρμογή. Τα στρώματα ε, συνομιλούν με άλλα αντίστοιχα στρώματα σε άλλα συστήματα. Έχουμε λοιπόν τον browser που μιλάει με έναν διακομιστή σε ένα άλλο σημείο. Ούτε ξέρετε, ούτε θέλετε να μάθετε πού. Η ανακοίνωση, η επικοινωνία μάλλον αυτή λέγεται in-to-in. -in, γιατί εσωτερική επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών. Αυτά τα στρώματα επίσης ε, έχουν επικοινωνία και με τα κατώτερα ε, στρώματα προέρχονται πολλές φορέ υπηρεσίε από το ίδιο το φυσικό μέσο μεταφορά. Βλέπετε πώς γίνεται αυτή η επικοινωνία, βλέπετε τις γραμμέ. Ε, γραμμές. Έχουμε δεξιά λοιπόν τον προσωπικό υπολογιστή και αριστερά έχουμε ένα διακομιστή, ένα σερβερ. Και στο μέσο θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφορα συστήματα, τα router που μεταφέρουν ε, την κυκλοφορία από το ένα σημείο του διαδικτύου στο άλλο μέχρι τον τελικό προορισμό. Ένα σημαντικό ερώτημα που έχει να κάνει την ουδετερότητα του δικτύου είναι όταν διαβιβάζουν την κυκλοφορία οι routers, πώς κάνουν, πώς ιεραρχούν τις προτεραιότητες. Και όταν σπάνια έχουμε υπερφόρτωση των γραμμών, τι θεωρείται επιτρεπτή συμπεριφορά σε αυτό το δίκτυο. Η απόδοση πολλά συστατικά. Πρώτα απ' όλα το εύρος της ζώνης. Πόσο μεγάλη είναι οι σωλήνε, δηλαδή, ποια είναι η δυναμικότητά του, πόσα beach ανά δευτερόλεπτο μπορούν να μεταφέρουν. Μία άλλη, ένα άλλο περιορισμό που δεν μπορεί κάνει να κάνει τίποτα και πολλά πράγματα γι' αυτόν είναι καθυστερήσει στη διάδοση, στη μετάδοση. Μήκος ε, του μεταμονοπατιού και ταχύτητα φωτό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτό. Επίσης, χρόνος αναμονής, ιδίως ε, στους ρούτερς μας από τους οποίους περνάει η κυκλοφορία και η καταπροτεραιότητα, ο καταπροτεραιότητα χειρισμός μπορεί να επηρεάσει αυτό το χρόνο αναμονής. Για τη συνολική απόδοση η μέση η καθυστέρηση έχει σημασία, αλλά και η ε, ποικιλότητα, αν θέλετε, η ποικιλομορφία αυτής της καθυστέρησης και τα δύο αυτά αλληλοεπιδρούν. Παραδείγματος χάρη, στη φωνητική ε, συνομιλία θέλουμε να υπάρχει ε, η αμφίδρομη αυτή μεταφορά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ενδιαφέρει λοιπόν και η ποικιλομορφία αλλά και ο μέσος όρο Και υπάρχει και το λεγόμενο packet loss, απώλεια πακέτων, που αυτά δηλαδή κάποια στιγμή κάπου πετιούνται. Το διαδίκτυο επιτρέπεται όταν είναι υποφορτωμένο, ε, είναι η κανονική συμπεριφορά, δεν είναι αστοχία. Αυτά λοιπόν ε, καθορίζουν τις αποδόσεις ε, του δικτύου. Είναι πράγματα όμως που βλέπουμε και εγώ ως προγραμματιστής, ως σχεδιαστής τα είδα, αλλά ως χρήστης μέρα δεν τα βλέπω. Ως χρήστες όμως ενδιαφερόμαστε όχι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά για το πώς αυτά επηρεάζουν την απόδοση και τις εφαρμογές. Η ποιότητα υπηρεσιών, οι παράμετροι αυτές που σας ανέφερα, είναι πολύ σημαντικές. Πώς επηρεάζουν όμως το χρήστη. Αυτό έχει να κάνει με το τι κάνουμε ω χρήστε. Κάποιε εφαρμογέ είναι πολύ ευαίσθητε, οι καθυστερήσει όλε άλλε όχι τόσο. Αν στέλνετε ένα email, η καθυστέρηση κάποιων δευτερολέπτων ή λεπτών μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία. Αλλά αν έχετε φωνητική επικοινωνία στο διαδίκτυο, φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 150 μιλισέκοντ να είναι διαφορά, η καθυστέρηση έχει πρόβλημα. Είχαμε 270 ε, μιλισέκοντ καθυστερήσεις όταν είχαμε δορυφορική επικοινωνία. Και τελικά μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Για το βίντεο, την οπτική επικοινωνία μπορεί να μην έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αν αν έχετε την καθυστέρηση των 2-3 δευτερόλεπτων στην αρχή ο χρήστη, ε, η ευαισθησία στην καθυστέρηση μετά είναι πολύ μικρή γιατί υπάρχει το λεγόμενο buffering στο σύστημα ε, υποδοχής. Δεν είναι πολύ σημαντική η καθυστέρηση. Επίσης το IPTV αν περιμένετε μισή ανταπόκριση όταν αλλάζετε κανάλι εκεί πάλι η καθυστέρηση είναι σημαντική. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν των επιδόσεων ε, του διαδικτύου εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση που κάνει ο χρήστη. Αυτά ό,τι το τεχνολογικό υπόβαθρο και α περάσουμε στο οικονομικό υπόβαθρο. Το οικονομικό υπόβαθρο τη ιδιαιτερότητα του δικτύου. Τρει βασικέ είναι οι συνιστώσει, θα έλεγα. Πρώτον, ποιοτική διαφοροποίηση. Δεύτερον, το λεγόμενο economic foreclosure, αποκάλυψη. Και δεύτερον, η διμερή ή δίπλευρη αγορά. Quality differentiation, ποιοτική διαφοροποίηση. Νομίζω όλοι το έχουμε ε, ακούσει. Πάμε σε ένα σταθμό ε, τρένων ή σε ένα αεροδρόμιο και μπορούμε να επιλέξουμε αν θα ταξιδέψουμε οικονομική ή πρώτη θέση. Και βέβαια υπάρχει διαφορά τιμών. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Εν γέννη, ε, στον οικονομολόγο αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση σημαίνει ότι αυτό βελτιώνει και την ευημερία του παραγωγού αλλά και την ευημερία του καταναλωτή. Δηλαδή αυτό θα σημαίνει ότι έχει περισσότερε επιλογές ο καταναλωτής. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί, ιδίω όταν υπάρχει ισχύ στην αγορά, με τρόπους που θα βλάψουν τελικά τον καταναλωτή. Το δεύτερο οικονομικό φαινόμενο είναι αυτή η οικονομική αποκάλυψη και είναι ένα από τα κύρια μελήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου. Ε, foreclosure είναι μία ε, έννοια ε, η οποία αφορά έναν παραγωγό ο οποίος δουλεύει στην αγορά και ο οποίος έχει την δυνατότητα να μεταφέρει σε ένα άλλο κομμάτι της αγοράς την ανταγωνιστικότητά του. Το παράδειγμα που δίνω εδώ είναι το εξής. είστε λοιπόν στον προσωπικό σας υπολογιστή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μηχανές αναζήτησης, Google ή Bing ή Yahoo ή οτιδήποτε άλλο. Ε, ε, βεβαίως, μέσω του δικού σας δικτύου, μέσω του δικτύου που σας δίνει ο πάροχός σας, θα περάσει ε, η μηχανή αυτή αναζήτησης. Εάν ο πάροχος ε, ευρυζωνικότητας έχει καλύτερη σχέση με έναν από τους πάροχους, τους παρόχους που ανέφερα προηγουμένως, ε, ενδεχομένως θα δυσκολέψει ε, για σας την πρόσβαση στους άλλους ε, παρόχους. Αλλά για φανταστείτε, ο ένας να θέλει να αγοράσει ή να εξαγοράσει τον άλλον. Ας πούμε η Yahoo να θέλει να εξαγοράσει τον τοπιο πάροχο ευρυζωνικότητας και αυτό θα το κάνει χρησιμοποιώντας και τη, δικιά σας παροχή. Και εάν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην υπηρεσία και το δίκτυο, ε, τότε θα μπορούσε να υπάρξει οικονομικό κίνητρο για να επιλέξει κανείς τον ένα ή τον άλλο πάροχο. Σημειώστε εδώ ότι η οικονομική δύναμη της αγοράς είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης αυτής. Εάν κάποιος προσπαθήσει να μπλοκάρει την ε, πρόσβασή μου σε ένα δίκτυο και αν έχω, ε, δίκ, ε, αν έχω ζημία από το κόστος καθυστέρησης ή αν έχω άρνηση πρόσβασης στο δίκτυο, τότε αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χάσει λόγω της συμπεριφοράς αυτής ο πάροχός μου ένα κομμάτι της αγοράς τη οικονομική θεώρηση. Είναι ένα νέο στοιχείο των οικονομικών. Ο, αλλά μπορεί να δει κανείς το ίντερνετ με τον τρόπο αυτό. Σε, σε μια δίπλευρη αγορά υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία συνδέει, μια πασαρέλα που συνδέει τις δύο πλευρές της ε, αγοράς. Ε, από τη μία πλευρά ας πούμε έχουμε ε, την ε, αναμετάδοση και από την άλλη μεριά έχουμε τον καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση οι διαφημιστές ε, ε, συνήθως είναι αυτοί που πληρώνουν ε, για τις υπηρεσίες. Κατά κανόνα οι καταναλωτές έχουν δωρεάν τις υπηρεσίες αυτές. Τώρα, σε μια αγορά για να έχει κανείς δωρεάν υπηρεσία ή κάτω του κόστους σε μια μονόπλευρη αγορά αυτό δεν γίνεται, είναι παράλογο, αλλά σε μια δίπλευρη αγορά είναι δυνατόν και φέρνει πολλές φορές κοντύτερα τη μία πλευρά της αγοράς με την άλλη και κάποιος πληρώνει, είτε από τη μία πλευρά της αγοράς είτε από την άλλη. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, λέω ότι είναι μια νέα οικονομική θεώρηση και είναι ένας λογικός τρόπος να δει κανείς το πρόβλημα αυτό. Ε, κατά αυτή την έννοια ε, τα προβλήματα τα οποία έχουν θυγεί σχετικά με την ουδετερότητα ενδεχομένως θα λυθούν εάν αντιμετωπίσουμε οικονομικά, με οικονομικούς όρους ε, το ερώτημα ποιος πρέπει να πληρώσει και γιατί πρέπει να πληρώσει η μία ή η άλλη πλευρά της αγοράς. Uh, Αυτό είναι το background. The next question is, how might that relate to business? Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι με ποιο τρόπο μπορούν να εξελιχθούν τα ε, ε, ε, business models. Νομίζω ότι είναι καλό να διαχωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν ενδεχομένως να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις. Ε, στο, ε, στο πρότυπο των δύο διαδρόμων του lane model έχουμε από τη μία μεριά ε, τον πάροχο ευρυζωνικότητας έχουμε δηλαδή μία, ένα διάδρομο ο οποίος θα αφορά το δημόσιο ίντερνετ με μεγάλες εξαιρέσεις την IPTV ας πούμε και επίσης ε, την μετάδοση φωνής ε, ε, μέσω του ίντερνετ. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν εύκολα να φανταστεί έναν κόσμο όπου το δημόσιο ίντερνετ συνυπάρχει στην ίδια ζώνη με το IP, την τηλεφωνία IP, το IPTV, την φωνητική μετάδοση και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια τάση η οποία καλύπτεται όλο και περισσότερο και πολλοί είναι οι πάροχοι οι οποίοι δουλεύουν με τον τρόπο αυτό. Συμβαίνει αυτό σήμερα λοιπόν. όμως αποτελεί προτεραιότητα ε, στη, ε, στον ενιαίο πάροχο. Εμείς ε, είδαμε τέσσερις διαφορετικές εξελίξεις του δικτύου. Στο, στη μία περίπτωση έχουμε ε, ε, αλλαγή, της, ε, αλλαγή των, του κόστους σε περίπτωση και επίσης συνέχεια και επιπλέον εξάπλωση του μοντέλου του Lane. Η άλλη δυνατότητα είναι ότι οι διάδρομοι οι οποίοι κατά προτεραιότητα χρησιμοποιούνται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους πάροχους. Ε, και ε, τέλος έχουμε τη δυνατότητα ε, του, της λεγόμενης υπηρεσίας end-to-end που δίνει την δυνατότητα, να, που δίνει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο δημόσιο ίντερνετ. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεχνικά μπορεί να γίνει και μπορούσε να γίνει εδώ και καιρό. Όμως δεν εφαρμόστηκε για μία σειρά οικονομικούς και εμπορικούς λόγους. και καλύπτονται βεβαίω στην ε, ε, έκθεση. Είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα για άλλους λόγους. Αυτό που προσπαθώ να δείξω με το γράφημα στην διαφάνεια αυτή ε, είναι ε, και ε, ο οικονομικός συσχετισμός των δυνατοτήτων και των μοντέλων που υπάρχουν. Αν τα δείτε προσεκτικά, θα δείτε ότι σε Business Managed IP και στο απλό IP έχουμε μία τάση μεγέθους και Κατά την άποψή μου, τα στοιχεία τα οποία είναι πιθανό να επαληθευτούν δίνουν ε, την δυνατότητα μια σχετική ε, αύξησης ε, και μια τάση που μπορούμε να την προβλέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Στα διάφορα σενάρια όμως βάζουμε άλλο input κάθε φορά. Περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια για να δούμε ότι τα σενάρια προφανώς ε, παρουσιάζουν ε, διαφορές ε, όσον αφορά και την επίπτωση που θα έχουν στον ανταγωνισμό. Όσον αφορά τώρα ακριβώς αυτό το θέμα της απειλής προς τον ανταγωνισμό, Νομίζουμε ότι το τρίτο σενάριο είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές Το, το τρίτο θα ήταν ίσως ε, το πιο ε, ε, δύσκολο, γιατί δεν είναι ανοιχτό στην, ε, στον ανταγωνισμό. Όσον αφορά το, το άνοιγμα του Managed IP Service, συγγνώμη, Service ε, Lane, ε, στην περίπτωση αυτή ε, έχουμε διαφορές επίπεδου και το ελεγχόμενο bitstream, η πρόσβαση ελεγχόμενη στην ροή των bit μπορεί να δημιουργήσει ενδεχομένως κάποια προβλήματα. Όμως το σενάριο το οποίο ενδεχομένω θα είναι πιο ελκυστικό για τους καταναλωτές είναι αυτό όπου υπάρχει ε, διασύνδεση ε, και επομένως άνοιγμα όλων των δικτύων. Ε, σας έχω ξαναπεί και το ξαναλέω ότι εδώ και 10-12 χρόνια είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο από τεχνική άποψη, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Uh, θα ήθελα να πω δύο κουβέντε σχετικά με τι διαφορές ανάμεσα στι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιστήσω προσοχή σας ε, στην διαφορετική δομή της αγοράς και τις ε, διαφορές που προκύπτουν από αυτό. Δεύτερον, διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο και τρίτον, διαφορετική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Η δομή της αγοράς λοιπόν είναι διαφορετική τα περισσότερα σπίτια στις ΗΠΑ μπορούν να έχουν ε, ευρυζωνικότητα είτε από την καλωδιακή τηλεόραση, από τον πάροχο τη καλωδιακή τηλεόραση, είτε από τον πάροχο των ε, τηλεπικοινωνιών. Ε, στην πρώτη περίπτωση έχουμε 38% ενώ το ADSL και το FTTH φτάνει περίπου στο 30% σύμφωνα με τα στοιχεία του FCC για το 2010. Το σύστημα είναι διαφορετικό λοιπόν ε, όσον αφορά τον πάροχο ε, καλωδιακής ευρυζωνικότητας. Οι ανταγωνιστικοί πάροχοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν είτε το LLU, είτε ε, μοιρασμένη πρόσβαση, είτε bitstream, έχουν περίπου εξαφανιστεί στις ΗΠΑ. Το μερίδιο της αγοράς τους δεν ξεπερνάει το 2%. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, ε, είχαμε δυνατότητες ε, εναλλακτικής ας πούμε ε, χρήσης αλλά ε, δεν υπάρχουν πλέον αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι το μερίδιο της αγοράς δεν ξεπερνάει το 2%. Το, το 2%. Όμως, στις ΗΠΑ ο ανταγωνισμός γίνεται ανάμεσα στους διαφορετικούς πάροχους καλλιδιακής ε, Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ε, η κινητή, ε, η ευρυζωνικότητα επί της κινητής ε, τηλεφωνίας και σε κινητά συστήματα, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα και όχι αντικατάσταση του σταθερού δικτύου. Δηλαδή πάντα, πάντα θέλουν την σταθερή ευρυζωνικότητα. Ας δούμε τώρα, τις διαφορε... Ας δούμε τώρα την διάθεση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη ε, η ανταγωνιστική δομή είναι πολύ πιο πλούσια. Ε, όμως ε, πρέπει να πούμε ότι είναι άνισα καταναμημένη η καλωδιακή κάλυψη στα κράτη-μέλη στις κάτω χώρες, στη Φλάνδρα, ε, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία έχουμε μεγάλη κάλυψη δικτύου, αλλά ε, στην Ιταλία ας πούμε το δίκτυο είναι πάρα πολύ μικρό. Η δεύτερη πολύ μεγάλη αγορά πάντως είναι ότι ε, το Shared Access, το LLU, το Bitstream αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του, του DSL που είναι η κύρια τεχνική της ευρυζωνικότητας. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βλέπετε λοιπόν ότι σε μερικές χώρες ε, υπάρχουν, υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ε, καταναλωτών ε, που δεν έχουν που δεν είναι γεγραμμένοι στον κεντρικό πάροχο αλλά στον ανταγωνισμό. Αυτές είναι, πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετικές αγορές με διαφορετική δομή. Το επόμενο σημείο τώρα, το κανονιστικό πλαίσιο. Βεβαίω το κανονιστικό πλαίσιο διέπεται και από τι διαφορέ τη αγορά. Στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουμε την έννοια που, την αντίληψη που έχει η Ευρώπη ότι υπάρχει ε, ε, ένας κεντρικός κανόνας που πρέπει να αφορά όλους. Στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες οι τηλεπικοινωνίες είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Στην πρώτη περίπτωση των τηλεπικοινωνιών που θεωρούνται ευαίσθητος τομέα, υπάρχουν πάρα πολλές κανονιστικές υποχρεώσεις. Αντιθέτως στην πληροφόρηση πάρα πολύ λίγες είναι οι υποχρεώσεις. τα τελευταία δέκα χρόνια ε, η, ε, η ευρυζωνική επικοινωνία ε, θεωρήθηκε υπηρεσία πληροφόρησης. Πράγμα που σημαίνει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια πολύ λίγα νομοθετήματα έχουν δημοσιευθεί όσον αφορά την μορφή αυτή τηλεπικοινωνίας. Τη στιγμή λοιπόν που η ουδετερότητα του δικτύου έγινε ε, ζήτημα ε, και άρχισε να συζητιέται, ε, οι Αμερικάνοι καταναλωτές ήταν λιγότερο καλυμμένοι, λιγότερο προστατευμένοι από τον ανταγωνισμό και αντιστοίχως λιγότερο προστατευμένοι από, τις, από ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Επομένως, το FCC των Ηνωμένων ε, θεώρησε ότι θα έπρεπε και το έκανε άλλωστε το Δεκέμβριο του 2010 να δημιουργήσει το λεγόμενο Open Internet Ruling. Ε, ε, και σε, αυτήν, σε, αυτόν τον, σε αυτό το νομοθέτημα βλέπουμε κανόνες οι οποίοι είναι γνωστοί ήδη στην Ευρώπη όσον και μάλιστα έχουν ήδη ενταχθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο του 2009. Έχουμε λοιπόν τον κανόνα που αφορά την διαφάνεια, έχουμε τον κανόνα που αφορά ε, την ε, μη... Ε, that I neglected to, to perhaps... τον μη αποκλεισμό, το no blocking ε, και επίσης τον κανόνα της ε, μη διακριτικής ε, μεταχείρισης. Όσον αφορά το δεύτερο κανόνα του no blocking, θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρχει blocking ούτε σε περίπτωση βίντεο, ούτε σε περίπτωση IPTV Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ε, σημείο γιατί ε, επανερχόμαστε σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως για την οικονομική αποκάλυψη στοιχείων. Ο τρίτος κανόνας ε, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία μη βάσιμη ή παράλογη διάκριση. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει ε, να δουλέψω λίγο για να δω τι σημαίνει ε, μη λογική ε, διακριτική μεταχείριση. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορετικά νομοθετήματα. Οι πρόνοιες για το LRU, Shared Access και Bitstream εξακολουθούν να είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματικές. Μέσω του άρθρου 8 της οδηγίας ε, ε, πλαίσιο αναφέρεται ότι ε, ε, ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο ε, κτλ. Ε, όλα διέπονται από ένα κανονιστικό πλαίσιο. Αναφέρεται σαφώς επίσης ότι θα, ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο, στις εφαρμογές, στις υπηρεσίες που επιλέγουν. Επίσης μέσα από διαφάνεια θα έχει την πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Ε, το, το θέμα του ανταγωνισμού ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ είναι μια άλλη ιστορία. Στις ΗΠΑ υπάρχουν ε, αποφάσεις δικαστηρίων πούμε που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ρύθμιση όσον αφορά την, τον ανταγωνισμό Ε, επομένως πρόκειται για μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να σας πω και φτάνω τώρα στα συστάσεις που θα αποτελέσουν και το κλείσιμο, το τέλος ε, της ε, παρέμβασής μου. Το σημαντικό είναι να, και αυτή είναι από τις κεντρικές μου προτάσεις, δεν πιστεύουμε ότι ε, πρέπει, ότι πρέπει να, ε, υπάρξει επιπλέον, να υπάρξουν επιπλέον υποχρεώσεις όσον αφορά ε, την ουδετερότητα του δικτύου. Ε, μέχρι ότου τουλάχιστον έχουμε αρκετά στοιχεία έτσι ώστε ε, να έχουν ε, αποδώσει καρπούσε οι υποχρεώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί μέσω των τροπολογιών του ρυθμιστικού πλαισίου του 2009. Επίσης ε, θα πρέπει να στηριχτεί και η τεχνική και η ε, πολιτική έρευνα, έτσι ώστε ε, να υπάρχει καλύτερη, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τους καταναλωτές. Τρίτον, πιστεύουμε ότι κάποιους από τους τομείς ε, ε, στους οποίους ε, έχουν αναφερθεί προβληματισμοί στη διάρκεια της διαβούλευσης όντως μπορεί να αποτελέσουν βάση συζήτησης και επομένως θα πρέπει περαιτέρω να μελετηθούν. Και άλλωστε αυτό κάνουμε. Όσον αφορά τα μελλοντικά βήματα, η φυσική ερώτηση είναι ε, τι θα κάνουμε εάν οι αποφάσεις που πήραμε το 2009 ε, δεν καρποφορήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντως να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος και πώς θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία βάσει των τροποποιήσεων του 2009. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ πληρή αυτή η παρουσίασή σας. και όπως είπατε και εσείς η, η δικιά μας επιτροπή ήταν υπεύθυνη για τα κύρια σημεία της ε, μεταρρύθμισης ιδίω και για τον στόχο της ε, διαφάνειας. <clears throat> και εισαγάγαμε και ορισμένα μέτρα που επιτρέπουν ε, να αλλάξουν τους προμηθευτές του κτίου οι καταναλωτές πολύ γλίγορα. Ιδίω ε, όσον αφορά το θέμα των ε, συμβάσεων μακρά διαρκείας που κατά βάση δεν επιτρέπουν στους ε, καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τι εξελίξεις της τεχνολογίας. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις για 10 λεπτά. Και καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονός ότι έχουμε δύο ομάδες ε, επισκεπτών, την ομάδα του Σίλαρα 20 επισκέπτες και του κυρίου Γκόρενς που μόλις έφτασε νομίζω. Εάν χρησιμοποιείτε λοιπόν το δίκτυο και πολλοί το χρησιμοποιούμε για facebook κλπ. Αυτές οι παρουσίες είναι για σας ιδιαίτερα και η υπεύθυνη πώς θα έρθει σε λίγο για να μας πείτε γιατί για το μέλλον. Θα το βρίσκετε πολύ ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος. Έχετε ερωτήσεις για τον παρουσιαστή όσον αφορά τα θέματα που παρουσίασαν. Μου φαίνεται ότι ο συνάδελφος που ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με το θέμα αυτό θα έχει κάποιες ερωτήσεις. Θα του δώσω το λόγο πρώτα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα και πολλές ερωτήσεις, λέει ο κύριος ε, Έξουρμ, γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ ε, σαφής. Κυρίως θα ήθελα να συμφωνήσω με κάτι που αναφέρεται μέσα στα πλαίσια της ε, πτυχής καινοτομίας που είναι τόσο σημαντική. Αυτό για μένα είναι το πιο κεντρικό θέμα. όταν μιλάμε για τα ελάχιστα πρότυπα, τι απαιτήσει που υπάρχουν. Ίσως έτσι λύσουμε κάπως ε, κάποια προβλήματα, αλλά το, τι θα είναι το μεγαλύτερο προσεχές ε, βήμα, το επόμενο Skype ας πούμε, θα είναι ελπίζω ευρωπαϊκό, κάποια μικρή εταιρεία στην Ευρώπη που δεν ξέρουμε καν θα το προωθήσει. Δηλαδή αυτό που ρωτάω είναι ότι εάν έχετε ε, μία μικρή εταιρεία startup που δεν έχει ε, καμία δυνατότητα δεν έχει κανένα πρόβλημα όσο δεν έχει επιτυχία. Όταν έχει επιτυχία όμως, ξαφνικά έρχονται οι τηλεφωνικές εταιρείες, τις χτυπάνε την πόρτα και τις λένε δεν θα ήταν πολύ κακό εάν ή ε, αρχίσετε να έχετε καθυστερήσει στο, στη χρησιμοποίηση του διαδικτύου κλπ. Υπάρχει δηλαδή αυτή, αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως. Γιατί υπάρχουν ε, καινούριε εταιρείε στην Ευρώπη τύπου Skype και έχουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που σας ανέφερα. Σχόλιο ήταν αυτό που είχα να πω, όχι ερώτηση. Πρόεδρος, ναι, ίσως είναι σημαντικό το σχόλιο σας, και θα τα συμπληρώσω, γιατί ένα από τα κέρια θέματα που θίγονται αυτή τη στιγμή και που σχετίζονται πάρα πολύ με την παρουσίαση αυτή που είχαμε είναι οι πτυχές των οικονομικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται. Εγώ θα ήθελα να πιέσω τον Μάρκο λίγο παραπάνω. Γιατί όπως μας έδειξε στις διάφορες πίνακες του, ορισμένες εταιρείες όπως η Google και οι άλλες, που πουλάνε τη διαφήμιση και έτσι είναι σε χαμηλό κόστος, λειτουργούν σε χαμηλό κόστος και μετά βασίζονται όμως στο να περάσουν οι διαφημίσεις αυτές στο, στους καταναλωτές. Και εκείνοι που επενδύουν εκεί ε, είναι πολύ ψηλού επίπεδου και αναρωτιόνται αν έχουν δικαίωμα σε ένα τμήμα αυτής της, ε, του, του εσόδου από τις διαφημίσεις. Παραδείγματος χάνει Skype. Η μεταφραση της φωνής απαιτεί υψηλό επίπεδο, επίπεδο ποιότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι μεταφορείς, αν πούμε έτσι, κυρίες, ε, χρειάζεται να έχουν ένα τμήμα των διαφημιστικών εσόδων για να μεταβάζουν πραγματικά το Skype. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει συνήθως η παρέμβαση όταν είναι πιο ενεργή η αγορά. Γιατί αυτά τα πολλά, πολλαπλά στρώματα στο οποίο αναφερθήκατε, ε, πώς να σας πω, σε μια πραγματικά ιδανικά αναγνωστική αγορά, ο καθένας σε κάθε στρώμα θα πρέπει να ωφελείται. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και θα πρέπει τις διακρίσεις να τις καταπολεμήσουμε. Ιδίω θα φροντίσουμε να υπάρχει αρκετό ανταγωνισμό. Αν κάποιο απορριφθεί δηλαδή από τη μία εταιρεία, θα μπορεί να πάει στην επόμενη. Και δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν ανταγωνιστική πρόκληση. Θα υπάρξει, όπω είπα, σήμερα σε μα διάταξη πριν να σας ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον Σκοτ Μάρκε για να απαντήσει, Ποιο άλλο θα ήθελε να υποβάλει ερωτήσει. σα αρκούσαν αυτά που ακούσατε φαντάζομαι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ακούσατε και εγώ είχαμε το, την ίδια παρατήρηση να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε. Πάρα πολύ ευφυή η ερώτησή σα. Καταρχήν οι ανησυχίε που εκφράσετε είναι νόμιμε. Δηλαδή, εάν το δίκτυο μπορεί να είναι Κατά κάποιον τρόπο ο φύλακα της πύλης ο θυρωρός και ελέγχει έτσι την αγορά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ίσως ορισμένες εταιρείες γι' αυτό ήδη έχουν εξαφανιστεί χωρίς να τις ε, πάρουμε καθόλου είδηση. το επιχειρήμα για, την, για το όφελος από την προσφορά των υπηρεσιών. Δεν είναι σωστό ότι δεν πληρώνονται αυτοί, αυτές οι εταιρείε, γιατί συνήθως πληρώνονται από την ε, υπηρεσία, από τον καταναλωτή. Και θα πρέπει να δούμε ότι μπορούμε επίσης να έχουν εισόδηματα από την άλλη πλευρά της αγοράς. Θυμάστε αυτά κάποιες διαφάνειες που που έδινε δύο προσφέροντε υπηρεσίε, ο ένα στον κατανοτή, ο άλλο στην ε, μηχανή αναζήτηση στο website. Αυτός που μου προσφέρει εμένα ε, την ευρυζωνική δυνατότητα δεν έχει ίσως άμεση άμεσο συμβόλαιο να δεσμευτεί για τον Google ή Yahoo. Όσον αφορά τώρα την πληρωμή για την ποιότητα και για το Skype, αυτό ήταν νομίζω το θέμα που έθιξαν πρώτοι οι, οι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καταναλωτών. Και οπωσδήποτε υπάρχει εδώ μια ανησυχία. Αν συζητάμε ότι αυτός που προσφέρει την ευρυζώνη, και θα επιβάλλει ένα τέλος στον καταναλωτή για τις υπηρεσίες αυτές, αυτό δεν νομίζω ότι θίγει θέματα ανταγωνισμού καθόλου. Είναι νομίζω λογικό το να ζητούνται περισσότερα χρήματα για πιο γλίγορη εξυπηρέτηση είναι φυσιολογικό. Εκεί που είναι πολύπλοκο είναι όταν θέλουν να επιβάλλουν τέλη και στην άλλη πλευρά της αγοράς. Πρόεδρος. Το άλλο που ενδιαφέρει στους πολλούς συναδέλφους και στο οποίο αναφερθήκατε είναι ότι είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις για το με Τελεκόμ όσον αφορά τις ε, παραβάσεις ε, του δικαιώματος, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Και υπάρχει κάποι, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουμε εισαγάγει εκεί. Η πρώτη περίπτωση στη ΣΥΠΑ ήταν νομίζω ότι κάποιοι είπαν ότι η επικοινωνία μεταξύ ίσων δεν είναι κάτι που δώσει το οποίο δώσουμε ολοκληρωτέ και γι' αυτό θα, θα το έχουμε πιο αργό για να δώσουμε τις πιο γρήγορες δυνατότητες σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν καλύψατε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας αξιολόγηση όμως πώς θα μπορούσε αυτό να προωθηθεί ίσως πολλοί από τους ακροτές μας εδώ πίσω, νομίζω πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε διαδίκτυο και διαφορώστε γι' αυτά, θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούν εκείνοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες να έχουν περισσότερη ευθύνη για το γεγονός ότι τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται και για παράνομα ε, σκοπούς. Εσεί πιστεύετε ότι μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα ή θα υπάρξει εδώ SAE στο διαδίκτυό μα. Νομίζω ότι εγώ προσπάθησα να τα κρατήσω εκτός έκθεσης αυτά, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, αλλά με πιάσατε στα πράσα όμως. Στη ΣΥΠΑ οι κανόνες λένε ότι κανείς μπορεί να λάβει το θεμητό περιεχόμενο, το νόμιμο περιεχόμενο. Εσείς λέτε ότι αυτό επειδή έχουμε άλλα τρία νομικά μέσα που το δεν χρειάζεται να το λέμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον όλη η κυκλοφορία peer-to-peer -peer είναι ειναι ό,τι αφορά δηλαδή το copyright. Υπάρχει και απόλυτα νόμιμη κυκλοφορία peer-to-peer. ΕΙΠΑ η Comcast, η εταιρεία, νομίζω ότι μετώπισε κάποια προβλήματα τα οποία σχετίζονταν με το ότι παρεμβαλόντουσαν με αυτή την κυκλοφορία peer-to-peer, αλλά ουσιαστικά μπλόκαραν την, ε, το upload και δεν κοινοποίησαν τους πελάτες τους ότι το έκαναν αυτό. Και αρχικά μάλιστα όταν ε, υπήρξαν τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο το αρνήθηκαν κιόλας Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία τίθενται και με τις διαφημίσεις και ίσως και να μην σχετίζονται πάντα μόνο με το copyright. Κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά δεν το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, αν ξεκινήσουμε με την αρχή ότι η ποιοτική διαφοροποίηση μπορεί να είναι θεμητή και νόμιμη αν ε, γίνεται για έγκυρους σκοπούς και με την ε, γνώση των καταναλωτών, τότε η, ε, το upload στο peer to -peer traffic μπορεί να είναι λιγότερο ε, σημαντικό και σε ό,τι αφορά το χρόνο, ε, παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα email ή σε σχέση με τη φωνητική τηλεφωνία στο πρωτοκόλλου διαδικτύου. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό είναι να μπλοκάρετε το uploading χωρίς να ενημερώνετε καταναλωτές. Σας ε, θέτω συνέχεια θέματα γιατί και οι άλλοι συνάδελφοι δεν φαίνεται να θέλουν να παρέμουν αλλά γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη η κυρία Κρούς. Και αφού είστε και εδώ, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας. Οπότε να σας ε, κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Επειδή έχουμε και πολλούς χρήστες του διαδικτύου εδώ στην αίθουσα. Μιλήσατε για τους ορισμούς της ουδετερότητας του δικτύου στην αρχή της παρουσίασής σας και είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι πιστεύουν ότι η ουδετερότητα δικτύου από την παρουσίασή σας ε, το αναφέρω, μιλά για την ίση μεταχείριση του περιεχομένου ανεξαρτήτως πηγής, ε, προέλευσης κτλ. η ισότιμη μεταχείριση αυτή της κυκλοφορίας ε, νομίζω ότι είναι θεωρητικό. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει συμβεί ποτέ στο διαδίκτυο αληθεύει νομίζω ότι το πρόβλημα που θα έχουμε στο μέλλον είναι ότι θα θέλουν να υπάρχει αυτή η μεταχείριση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Άρα θα χρειάζεται και η σχετική νομοθεσία. Ποια είναι η δική σας άποψη. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να μας ε, σχολιάσετε. Αυτό που για μένα είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα. και μας ζητούν να το κάνουμε αυτό ως νομοθέτες. Απάντηση. Και από τεχνική από οικονομική πλευρά νομίζω ότι ο δεύτερος ορισμός ε, δεν είναι σωστή ιδέα. Υπάρχουν οικονομικά επιχειρήματα, ευσταθεί ότι ε, πράγματι πρέπει να γίνεται κάποια διαφοροποίηση ποιότητας, αλλά να μην σχετίζεται βέβαια με διακριτική μεταχείριση που θα μπορεί να βλάψει τον ανταγωνισμό. Υπήρξαν βέβαια επιχειρήματα και στη βιβλιογραφία και στον τύπο που υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο πάντοτε προσχωρεί στις λεγόμενες αρχές in-to-in ε, και δεν κάνει καμία ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Αυτοί όμως αγνοούν την ιστορία, αγνοούν το παρελθόν. Σε ερευνητικό τώρα επίπεδο, σε επίπεδο έρευνας, η προτεραιότητα είναι μέσα στις ίδιες προδιαγραφές του διαδικτύου, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν το 1981. Και αν πάτε πίσω ε, στο OpenNet, που είναι ο προκάτοχος ε, του διαδικτύου, είχα εργαστεί για μια από αυτές τις εταιρείες το 69, την BBN, η πηγαίνουμε πίσω στο 73 και την έρευνα που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ε, για την ποιότητα της υπηρεσίας η ποιότητα της υπηρεσίας υπάρχει. Και φυσικά ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους στρατιωτικούς. Η εταιρεία μου μετέφερε κατά προτεραιότητα φωνητικά μηνύματα στη δεκαετία του 80 για τους ε, στρατιωτικούς και στη δεκαετία του 90. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη προϊστορία ιεράρχης προτεραιοτήτων Μην πάμε λοιπόν να ξαναγράψουμε την ιστορία. Τώρα από οικονομικής πλευράς νομίζω ότι επίσης υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα που συνηγορούν στο ότι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων ε, έχει τη σημασία της για κάποια είδη κυκλοφορία, αλλά δεν θα πρέπει να είναι διακριτική. Τότε μπορούμε να τη δεχθούμε. Αν συνιστά μεταχείριση, διακριτική μεταχείριση όχι. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. Εγώ ενδιαφέρομαι, αλλά φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι. Μπορείτε λοιπόν ε, να πάρετε αντίγραφα, μόλις έδωσε ένα αντίγραφο στην Επίτροπο, που ίσως θέλει να το μελετήσει το Σαββατοκύριακο, Ω ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. Όπως έλεγα κυρία Επίτροπε, όπως προβλέπει, όπως ε, μάλλον ε, συμπεραίνει και η μελέτη, νομίζω ότι έχουμε και τη διάσκεψη κορυφή τη εταιρεότητα του δικτύου πρόσφατα. Νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν σε αυτά τα οποία ε, υποστηρίζετε και εσείς. Ε, θα μας πείτε στο πρόγραμμα εργασίας σας τα σχετικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σκότ Μάρκους και νομίζω ότι το αξίζει χειροκρότημα παρακαλώ του κυρίου Μάρκους. Uh, uh, uh, Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να περάσουμε ευθύ αμέσω ε, στην Επίτροπο, την αρμόδιο για τα θέματα της ψηφιακής ατζέντα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας κύριε Κρούς. Συζητήσαμε διάφορα θέματα με τους επιτρόπους. Είχαμε υποδεχθεί τον κύριο Σέμετα, τον κύριο Ντάλι, μιλήσαμε για τα δικά τους προγράμματα εργασίας. Και τώρα έχουμε εσάς, έχουμε ένα αντίγραφο των βασικών πρωτοβουλειών για τις οποίες θα μας μιλήσετε και έτσι θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι βουλευτές. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν καταρχάς να μας παρουσιάσετε τις ιδέες σας και στη συνέχεια να δεχθείτε ερωτήσεις από τους συναδέλφους βουλευτές. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας. Νιώθω ότι πραγματικά μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Μπορώ και εγώ πράγματι κάποιες από τις παρατηρήσεις σας ε, να τις ε, ε, χρησιμοποιήσω σε λαβή για σκέψη, τροφή για σκέψη. Και να σας πω ότι χθες στο Παρίσι είχα μια πολύ συναρπαστική ε, συνάντηση στο πλαίσιο του G8 και η Κομισιόν αλλά και κάποια, μέλη του, κάποια κράτη-μέλη δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το διαδίκτυο και την ψηφιακή οικονομία. Όπως ο πρώτος Σαρκοζή για παράδειγμα, που προείδρευσε της ομάδας των 8 και ανέφερε το θέμα αυτό της ψηφιακής οικονομίας ως προτεραιότητα. Κάθε μέρα στις 27 χώρες μέλη έχουμε συνεργασία και με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς για να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία. Εκεί εντάσσεται και η λεγόμενη ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο. πολλοί που παίρνουν από τις Βρυξέλλες έχουν συναντήσεις και με εσά ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά όλα αυτά δείχνουν πόσο πολύ ε, ενδιαφέρον υπάρχει για αυτό το θέμα. Όταν μιλάμε μάλιστα για μια τεράστια αλλαγή στην κοινωνία των πολιτών, μια τεράστια αλλαγή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας Πολύ σημαντική λοιπόν η στιγμή αυτή, χωρίς καμία αμφιβολία, για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, διότι οι αναθεωρημένοι κανόνες τέθησαν πλέον σε ισχύ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Επιτροπή σας, διότι βοήθησε στην ε, διαμόρφωση ενός βελτιωμένου ρυθμιστικού πλαισίου που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη συνέχεια ε, στις αργές ε, στις οποίες βασίστηκε, αλλά συγχρόνως και για τον καθορισμό νέων διατάξεων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πολλές μελλοντικέ προκλήσεις. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας τώρα είναι να παρακολουθήσουμε την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών αυτής της αναθεωρημένης, ε, του αναθεωρημένου τηλεπικοινωνιακού πλαισίου. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της ετήσια έκθεσης για την πρόοδο της ε, αγοράς τηλεπικοινωνιών. Μετά την έγκριση του ψηφιακού θεματολογίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσαρμόσει την παραδοσιακή της δομή υποβολής εκθέσεων για την 16η επικείμενη έκθεση πρόοδου και να εκδώσει το λεγόμενο scoreboard, ε, τον πίνακα επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου. Ο στόχος είναι να έχουν ε, στοιχεία συγκεκριμένα, νούμερα συγκεκριμένα τα έγγραφα αυτά. Δύο τον αριθμό θα δημοσιευθούν στα τέλη του μήνα. Μέχρι στιγμής μόνο τρία έχουν ολοκληρώσει όλα τα βήματα για την πλήρη υλοποίηση του πλαισίου. Τα περισσότερα κοντεύουν να τα ολοκληρώσουν, αλλά υπάρχουν και ορισμένα τα οποία δυστυχώς είναι πολύ πίσω. Τέσσερα συγκεκριμένα είναι πολύ πίσω. Βέβαια, δεν θα διστάσουμε να κινήσουμε και διαδικασίες επί παραβάση για τη μη συμμόρφωση, εάν δεν μεταφερθεί γρήγορα το πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο. Προς το παρόν απλά το λέμε ώστε να προσπαθήσουν οι τέσσερις κακοί μαθητέ, οι τέσσερις ουραγοί, να σημειώσουν την τραπετούμενη πρόοδο για να φτάσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ξέρετε επίσης ότι πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία ανακοίνωση για την ουδετερότητα δικτύου. Έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις, υπήρξε και μία διάσκεψη Κοινοβουλίου Επιτροπής και εσεί ω ε, Επιτροπή διδραματίσετε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την διάσκεψη. Και όλα αυτά τα απορίσματα τα συμπεριλάβαμε σε αυτή την ανακοίνωση θα φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια, ποιότητα υπηρεσίας και δυνατότητα αλλαγή ε, παρόχου με τους νέους τηλεπικοινωνιακούς ε, κανόνες. Και βέβαια όλα αυτά κατά τρόπο ώστε να υπάρχει σεβασμός ε, στις, ανοιχτές, στις αρχές περί ανοίγματος και περί ουδέτερου διαδικτύου. Η ομάδα των Ευρωπαίων Ρυθμιστικών Αρχών η Μπέρεκ, εκλήθη επίσης ε, να προβεί σε μια διευνητική αποστολή για θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για ένα ανοιχτό και ουδέτερο διαδίκτυο. Παραδείγματο χάρη εμπόδια για την αλλαγή παρόχου ή η παρεμπόδιση ή ο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο φωνητική παραδείγματος χάρη μετάδοση σε βάρος των διαδικτυακών υπηρεσιών, διαφάνεια, ποιότητα υπηρεσιών. Στα τέλη του χρόνου, αφού έχουμε τα στοιχεία μας ε, της ε, Μπέρικ, θα τα δημοσιεύσουμε και αν χρειαστεί θα προβούμε και στην έκδοση περαιτέρω καθοδηγητικό, καθοδη, ε, κατευθυντηρίων γραμμών, ίσως και νομοθετικών πρωτοβουλειών. Τώρα, η καθολική υπηρεσία στο πλαίσιο τη ευρυζωνικότητα ήταν ένα ε, θέμα δημόσια διαβούλευση πέρυσι. Είναι επίση ε, σημαντικό το θέμα αυτό και εκεί πρέπει να καταφέρουμε να εξισορροπήσουμε με πολύ προσεκτικό τρόπο τα διάφορα ε, πολύ σημαντικά δημόσια συμφέροντα. Το σχέδιο έκθεση επιτροπή σα για την καθολική υπηρεσία και για τον αριθμό τη ανάγκη το 112, χθε νομίζω το ψηφίσατε, νομίζω ότι βοηθάνε στο να έχουμε αυτή την πολύ καλή ισορροπία. Αργότερα φέτος ε, θα αναφέρω στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με την έκβαση της δημόσιας διαβούλευση και θα σας πω πώς βλέπουμε εμείς την εφαρμογή των ρόλων της Ένωσης ό,τι αφορά την καθολική υπηρεσία στο ευρυζωνικό περιβάλλον. Έρχομαι ε, σύντομα στο νούμερο 112. Το αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύει σημαντικά τις υποχρεώσεις ε, για τις υπηρεσίες ε, έκτακτης ανάγκης για τον αριθμό 112. Έχουμε ενισχύσει τις υποχρεώσεις ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ε, ισότιμο, ισοδύναμο με όλους τους άλλους χρήστες επίπεδο πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να πω επίσης ότι η τεχνική πρόοδος θα είναι πολύ μικρή εάν δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Πώς να χρησιμοποιήσεις μια υπηρεσία που δεν ξέρεις ότι υπάρχει. Άρα το πρώτο βήμα είναι αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι ένας στους τέσσερις πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα γνωρίζει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στο 112 όλες ε, τις ώρες της ημέρας, 24 ώρου βάσεως και σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για οποιαδήποτε, ε, περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Είναι σοκαριστικό αυτό το νούμερο, Ένα στους 4. Πρέπει να αλλάξει αυτό, δεν μπορούμε να παίζουμε με την ανθρώπινη ζωή. Να αναφερθώ επίσης συντομία στο e-call, μια υπηρεσία λοιπόν ηλεκτρονικών κλήσεων διαλειτουργική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον αριθμό έκτακτη ανάγκη 112 η εισαγωγή αυτής της υπηρεσίας θεωρούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα βραχυχρόνια μέτρα για να μειώσουμε τα μοιραία ε, τροχαία δυστυχήματα και τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Μεγάλη προτεραιότητα για την Κομισιόν και σύντομα θα υιοθετήσουμε σύσταση προς τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών κλήσεων. Θα είναι το πρώτο, τα τρία νομοθετικά μέτρα που θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση του e-call σε όλα τα οχήματα που έχουν τη νέα έγκριση τύπου, δηλαδή από το 2015 και μετά. Επίσης, ένα θέμα που φαντάζομαι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η περιαγωγή. Είναι σημαντική η περιαγωγή, είναι σημαντική για τους επιχειρηματίες, για τους ε, τουρίστες και βέβαια κυρίως για όσους ε, προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά αποφασιστικά προς το κοινό όφελος και προς το κοινό συμφέρον. Έχουμε τους τρέχοντες κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά το πρόβλημα το ουσιώδες δεν έχει αντιμετωπιστεί. Θέλουμε δηλαδή να υπάρξει μείωση των τιμών λιανικής και καλύτερος ανταγωνισμός, ιδίως για τα δεδομένα. Πρέπει ε, επίσης ε, να λύσουμε τα ζητήματα του υποκείμενου ανταγωνισμού. Έχει αποτύχει αγορά μέχρι στιγμής και εγώ πρέπει να σας πω ότι σκέφτομαι μια υβριδική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διαρθρωτικά στοιχεία, δομικά στοιχεία που θα προωθούν την είσοδο στην αγορά και θα βελτιώνουν το φάσμα επιλογής του καταναλωτή για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Θα πρέπει επίσης να είναι σταθερό. Θα πρέπει να έχει ασφαλιστικές δικλείδες μέχρι ότου μπορέσουν να ισχύσουν πλήρως τα δομικά ενδικά μέσα. Ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχει εγκριθεί η πρόταση. Τουλάχιστον θα είναι έτοιμη μέχρι τότε. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή σας και την Προεδρία για την υποστήριξή σας ε, με την γνωμονότητα που δώσετε στην Επιτροπή ΙΤΡΕ για την ε, στρατηγική ευρωζωνής της ε, Κομισιόν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει οι καταναλωτέ να στο επίκεντρο των προσπαθειών μα για να φτάσουμε εκεί. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερε ε, περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις όπως το Project Bonds Initiative που παρουσιάζει στις 8 Φεβρουαρίου και ένα νέο μέτρο για τη, τα δίκτυα του μέλλοντος στις μεταφορές ενέργεια και ICT και ε, Ευρωζωνία. Όλοι υποστηρίζουν με την ιδέα αυτή. Θα είναι λοιπόν, ε, θα περάσει από την επίσημη διαδικασία λήψη απόφαση ε, του Συλλογικού Οργάνου της Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να υπάρχει σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που θα καλύψει μέχρι το 2020 ένα μεγάλο ποσοστό του χάσματος για τη χρηματοδότηση της Ευρωζώνης. Βέβαια, η συμβολή της Ευρώπης είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των ε, υπηρεσιών αυτών ε, της, ε, του ICT. Τα ωφέλη πολλαπλασιάζονται και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις υπηρεσίες της, του e-government, του ηλεκτρονικού, της ελληνικής κυβέρνησης που δίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δίνει τη δυνατότητα δράση στου πολίτε και στι επιχειρήσεις. Γι' αυτό το προγραμμα δραση δράσης 2011-2015 που έχει σαν στόχο ο δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ευέλικτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί ενδυναμώνει και την ενιαία αγορά. Η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς οπωσδήποτε έχει σαν στόχο να αυξήσει την εσωτερική ζήτηση και να καταστήσει την οικονομία πιο ανταγωνιστική πλήρως ισομετωμένη αγορά για ηλεκτρονικό εμπόριο είναι στο επίκεντρο του οράματο αυτού. Και γι' αυτό θα σα ευχαριστώ για τη συμβολή που έλαβα από την ομάδα εργασία IMCO για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το e-commerce. Μελέτησα την, ε, έκθεση που προετοιμάσατε, που οδήγησε στο ψήφισμα του 21 Σεπτεμβρίου 2010 και πιστεύω ότι είναι απόλυτα ευθυνασμένη με τις ε, φιλοδοξίες της ε, ψηφιακή, του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Θα λάβω υπόψη μου αυτή την συμβολή σας για την προετοιμασία της ψηφιακής ατζέντα για το ψηφιακό θεματολόγιο, δηλαδή μέχρι το έτη του 2012. Ε, επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι η, το θέμα του e-health, ηλεκτρονική υγεία, που αφορά και ενδιαφέρει άμεσα τους πολίτες. Παραδειγματικά, θα ήθελα να σας πω ότι θέλω να υποβάλω προτάσεις για μέτρα μέχρι το 2012 όσον αφορά ένα ελάχιστο επίπεδο στοιχείων των ε, ασθενών και έτσι θα μπορεί το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό μιας χώρας να έχει στοιχεία για την υγεία κάποιου ασθενούς που έπαθε παραδείγματος ένα δυστύχημα ή αρρώστησε εκτός της χώρας του. Και επίσης προωθώ ένα σχέδιο Active and Healthy Aging, υγιή και ενεργή μεγάλη ηλικία που προωθεί τη χρήση της τεχνολογίας για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων τόμων και εκείνων που τους περιθάλπτουν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα παρακολούθησης χρονίων ασθενειών, πρόληψη και ε, τεχνολογίες υποστήριξης. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τομέα της υγείας και ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμο στο εγγύς μέλλον για οποιοδήποτε. Παρ' αυτά ακόμα πρέπει πολύ να προχωρήσουμε για να προωθήσουμε τη χρήση των υπηρεσιών online. Οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς να χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες και οι αρχές και οι υπηρεσίες θα πρέπει επιχειρήσεις να τις αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό, όπως το ίδιο το Ιντερνετ, το διαδίκτυο θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και διασυνοριακά. Και γι' αυτό θα πρέπει και ο δημόσιος και ο τομέα να δούμε ότι ζητούν σήμερα μια ηλεκτρονική ταυτότητα για να μπορεί να υπάρχει ασφαλής ε, ε, προσβασή στις υπηρεσίες τους αυτές online όμως μέχρι στιγμή ε, σταματάνε στα σύνορα ενώ θα έπρεπε να λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό θέλω να προτείνουμε μια νομική βάση για τα κράτη-μέλη να δέχονται τις αυτότητες και από τις άλλες ε, ε χώρες μέλη. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 450 απαντήσεις στην διαβούλευση που κάνουμε για το θέμα και θα συνεχίσουμε μέχρι την σύνοδο της, του ψυχιακού θεματολογίου τον Ιούνιο. Ελπίζω ότι πολλοί από εσά θα μπορούν να είναι παρόντες σε αυτή την εκδήλωση γιατί θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανταλλαγής σκέψεων αλλά και συγκεκριμένων προτάσεων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Ξέρω ότι πολλοί από εσά ήδη έχουν ε, δεσμευτεί και ασχολούνται με αυτό την εκδήλωση που θα κινητοποιήσει το θέμα των ε, ταυτοτήτων για τις ε, νέες μας δράσεις. Επίσης ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της προσδετώτης πρόσβασης στο δίκτυο Web Accessibility. Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούν αυτές οι, αυτές οι να είναι πλήρως προσβάσιμες μέχρι το 2015. Και για να το πετύχουμε αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή μία αξιολόγηση των επιπτώσεων για να δούμε ποια θα ήταν η καλύτερη πολιτική δράση, ενδεχομένως και νομοθεσία, που θα μπορούσε να βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσματική και δανεισμένη η εφαρμογή αυτής της προσβατότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Κομισιόν θα προωθήσει τις προσπάθειές της για πολλούς τομείς νομοθεσίας, ανάπτυξη και απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ποιότητα ζωής, μαζί με τα σχέδια μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για να μπορέσουμε έτσι να σεβαστούμε και την Σύμβαση των, Ανθρωπίνων, των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβατό σε όλου όπω θα έπρεπε, αλλά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό. Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι όλοι ανησυχούμε για τι απειλέ στην ε, ασφάλεια στον κυβερνόχωρο. Όλοι ε, αναλαμβάνουμε πράξεις ε, για να το προωθήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέρα από αυτό. Έχουμε εδώ τις νομοθετικέ προσπάθειες τη ΕΝΙΣΑ που θα αυξήσει τις δυνατότητες και θα βελτιώσει τις ε, λειτουργίες της. Επίσης συνεργαζόμαστε σε με κράτη-μέλη για να προχωρήσουμε και να επιταχύνουμε την εφαρμογή του προγράμματος δράσης ε, για τις κρίσιμες πληροφορίες για την προστασία των υποδομών. Επίσης έχουμε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας της ΕΠΑ σαν τμήμα μιας ομάδας εργασίας που ασχολείται ακριβώς με το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνόχωρο και τα εγκλήματα στον κυβερνόχωρο. Είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον ε, εταίρο μου από αμερικανικής πλευράς και επίσης είναι άδελφος σε Σίλια Μάρσον στην Κομισιόν και η είχαμε αυτή τη συνάντηση και θέλαμε και οι δύο να καταλήξουμε γλίγορα σε συγκεκριμένη μέτρα και ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε αυτό μέχρι τον Νοέμβριο. Να υπάρχει δηλαδή μια, ένας κατάλογος αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ε, τυποποίησης. Πολλά σημαντικά πρότυπα χρησιμοποιούνται σήμερα σε κάθε ε, σχετίζεται με το διαδίκτυο, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό τι σημαίνει. Δεν έχουν εκδοθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης. Και αναφέρομαι σε διάφορα πρότυπα για φόρα που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ε, οργανώσεις. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα ε, πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιούνται πολύ καλά και στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως σημαντικά για την αγορά ICT όλα τα πρότυπα αυτά και δεν λειτουργούν όλα διαφανώς και γι' αυτό η μεταρρύθμιση της υποποίησης θα εγγυώται ότι τα πρότυπα που επιλέγονται για τις δημόσιες προμήθειες και την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ασφαλή ε, πρότυπα. Η πρόταση για τη με τη νομοθεσία τυποποίηση θα υποβληθεί σύντομα από την Κομισιόν. Αυτά θα είναι τα στάνταρ, που, τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία και καλύπτουν το σημερινό διαδίκτυο. Και θα ορίζουν πώς θα είναι το διαδίκτυο του την αύριον ή στο μέλλον. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι καυτό το θέμα του cloud computing και το Internet of Things. Είναι πολύ ελκυστικό. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις και ανοίξαμε μία δημόσια ε, διαβούλευση για να έχουμε μία νομοθεσία για την Ευρώπη ούτως ώστε όλοι όσοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με το θέμα να μπορέσουν να μας δώσουν κάποιες ιδέες, κάνουν κάποιες προτάσεις. Δεν πρέπει να κάνω εγώ τη δουλειά τους και εκείνη τη δική μου δουλειά, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας παρουσιάσουν πρωτοβουλίες, να παρουσιάσουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή και να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Η επόμενη, η επόμενη <clears throat> γενιά, ιδίω μέσω του Internet of Things και του Cloud Computing, θα πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα για τη συλλογή στοιχείων, ανταλλαγή, επεξεργασία και τα συστήματα θα μπορούν μάλιστα να κάνουν και αυτόματες αποφάσεις. Η χρήση των συστημάτων και των στοιχείων θα μπορούν να μας προσφέρουν μια πιο πράσινη και καλύτερη κοινωνία, αλλά όχι εάν οι πολίτες νομίζουν ότι δημιουργούμε εδώ έναν εφιάλτη, όπως αυτό που παρουσιάζει ο Όρβελ το 1984. Λόγω του ότι τα πράγματα είναι τόσο αλληλοσυνδεόμενα, δεν μπορούμε πάντα να εξασφαλίζουμε ίσως την ιδιωτική τομή. Θα πρέπει η, η προστασία της ιδιωτικής ζωής να, έχει, ε, να είναι ένα αναπόσπατο τμήμα κατά το συνδυασμό των συστημάτων αυτών. Θα πρέπει να υπάρχουν λύσεις λογισμικού που θα μπορούν οι ε, πολίτες να αποσυνδεθούν προσωρινά ή οριστικά από το δίκτυο. Αυτές οι ιδέες και άλλες πολλές συζητιούνται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογνωμόνων για το πρόγραμμα αυτό Internet of Things που ξεκίνησα πέρσι. Πρόκειται για ένα μακρύ κατάλογο απλώς σας λέμε τι κάναμε, τι κάνουμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις παρεμβάσεις, τα σχόλιά σας, τις ε, επικοδομητικές σας ιδέες για αυτό τόσο ευρύ θέμα. Και με ενδιαφέρον θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε για πολύ, τις πολύ σαφείς και πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στις οποίες αναφερθήκατε. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας εδώ ε, παρακολουθεί όλα αυτά τα, ε, τα σημεία σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει για την προστασία των καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς. Ε, πραγματικά θέλουμε ε, να δούμε τα, τον νέο κατάλογο των δικαιωμάτων των ε, χριστών Η οδηγία για τα, δικαιώματα των χριστών ήταν ένα δικό μας παιδί και πραγματικά περιμένουμε με μεγάλη προσδοκία να δούμε τι πρόκειται να γίνει στον τομέα αυτό. Θέλουμε ε, το Digital Scoreboard, το, το δικτυακό βαθμολόγιο να ε, ε, προωθηθεί και βεβαίως να λάβει υπόψη κάποια πολύ κεντρικά σημεία όπως είναι η διαφάνεια, όπως είναι οι συμβάσεις, όπως είναι η δυνατότητα αλλαγής παρόχου, διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά κατά την άποψή μου. Ε, θα δώσω μετά από μένα τον ε, λόγο στους εισηγητές που δουλεύουν πάνω σε ε, σχέδια τα οποία αφορούν την τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ο κύριος Αρίας, ο οποίος δουλεύει για το θέμα της ψηφιακής ενίας αγοράς, ο κύριος Ροσφόρ για το θέμα της επίλυσης διαφορών. Βεβαίως θέματα που αφορούν την προστασία των πολιτών ή στην κυρία Αράπτη ε, η οποία χθε παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ε, μια έκθεση στην Επιτροπή μας ε, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή. Είναι θέματα τα οποία λοιπόν απασχολούν την, έκθεση, την Επιτροπή μας. Συγγνώμη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους προαναφερόμενους και μετά έχω άλλους συγγεγραμμένους, την κυρία Βάλη και άλλους δύο. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν. Ε, κύριος Αρίας πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρέα στην παρουσίασή σας ε, και για την ηγετική στάση που δείχνετε σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή που ζούμε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πάω στην ομάδα εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΙΜΣΟ έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά ε, και έχει εμπλουτίσει τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας μας ε, που καλό θα ήταν ίσως αν μπορέσετε να έρθετε κάποια στιγμή και σας ευχαριστούμε πάντως για όσα κάνετε. Σε ό,τι αφορά το EG8, το φόρουμ αυτό στο οποίο μας αναφέρατε και στο οποίο πήγατε και στη Γαλλία, ε, πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία, πολύ ενδιαφέρουσα. Και όπως είπατε και χθε, πράγματι και εγώ πιστεύω ότι το δίκτυο απαιτεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες του παιχνιδιού, που θα είναι παγκόσμιοι. Διότι το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο, δεν είναι κάτι τοπικό, δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Οι κανόνες Είπατε ότι θα πρέπει να είναι κανόνες που θα αποτρέπουν το, την παράνομη μεταμόρφωση, μεταφόρτωση συγγνώμη, ε, περιεχομένου. Επίσης, ανάγκη να εκπαιδεύσουμε ε, ήδη από νεαρή ηλικία ε, τα παιδιά σε αυτή την ψηφιακή τεχνολογία, για την ψηφιακή εποχή, που θα πρέπει να μαθαίνουν να κάνουν καλή χρήση των νέων τεχνολογιών. Και αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ίσως και στο πλαίσιο αυτών των παγκόσμιων κανόνων. η Κομισιόν εγκρίνει κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την εκπαίδευση από την ε, μικρή ε, παιδική ηλικία και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Ε, Κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ο Μάλκολμ Χάρμπορ αναφέρθηκε στο σύστημα των online dispute resolution, επίλυση ε, διαφορών ε, για το διαδίκτυο, για τις επιγραμμικές υπηρεσίες ε, όσον αφορά τις απλές μη επιγραμμικές δηλαδή επιλύσεις διαφορών έχουμε ήδη προχωρήσει αλλά όσον αφορά τις online διαδικασίες έχουμε μείνει πολύ πίσω στην ε, πράξη για την ε, νέα αγορά λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο αυτό. Όμως λέγω ότι οι δύο πρωτοβουλίες θα πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό διασύνδεσης, γιατί τελικά αυτό που ενδιαφέρει τους καταναλωτές πολίτες είναι να λυθεί το πρόβλημά τους έστω και εάν έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετική τεχνολογία ή μέσο για να αγοράσουν το αγαθό όσον αφορά την δημοσίευση ε, του κώδικα των δικαιωμάτων ε, για τις ε, αγορές online. Μας είπατε 2012, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι να είναι ορατός, να είναι γνωστός αυτός ο κώδικας, γιατί δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιά τους και τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές. Τι θα κάνετε λοιπόν έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι διαδικασίες αυτές. Ξέρουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές και στο ε, e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο ε, και σε όλες τις επιγραμμικές ε, διαδικασίες. Επομένως, ανάλογα με τα, διάφορα τομεακά ενδιαφέροντα, θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος αντίστοιχος των δικαιωμάτων των καταναλωτών, αλλά και των δικαιωμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές αυτές οι ιδέες. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Ε, κυρία Κρός, με πάρα πολύ χαρά άκουσα την τοποθέτησή σας ειδικότερα για το θέμα του Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 ε, για το οποίο το είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Είχαμε χθες, ψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή μας μια έκθεση. Θέλω να σας ενημερώσω και το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ότι η έκθεση αυτή έγινε με πολλή δουλειά και με μια εξαιρετική συνεργασία όλων των σκιωδών συναδέλφων από όλες τις πολιτικές ομάδες, όλων των άλλων συναδέλφων που ε, πάρα πολύ εργάστηκαν και φρόντισαν για την έκθεση και πρέπει δεν να σας πω ότι ήταν πολύ έντονη και η παρουσία και της γραμματείας και των βοηθών όλων μας. Τα λέω όλα αυτά για να γίνει απολύτως σαφές το πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η υπόθεση του 112 και της καθολικής υπηρεσίας. Ήταν μια υπόθεση που μας άγγιξε όλους. Καθώς λοιπόν είμαστε στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, ε, θα ήθελα να ακούσω, έχοντας και τη δική μας στήριξη, τι πια προτίθεστε να κάνετε με περισσότερη λεπτομέρεια για να προχωρήσουμε. Και μία μικρή ερώτηση που αφορά τον ΕΝΙΣΑ. Πάω σε ένα άλλο θέμα, την ασφάλεια των δικτύων. Και σκέπτομαι, ε, εργαζόμαστε για την ασφάλεια των δικτύων. Μήπως πρέπει να εργαστούμε και για την ασφάλεια εντός εισαγωγικών αυτού ακριβώς του οργανισμού του ΕΝΙΣΑ, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δέχεται κάποιες επιθέσεις. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από την Επίτροπο κ. Νελικρούς να απαντήσει σε αυτή την πρώτη σειρά των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, και ευχαριστώ και κύριε εισηγητά ε, Χάρμπορ. Πραγματικά ε, είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένη και ευγνώμων για την εργασία που κάνουν οι εισηγητές και οι σκιώδες εισηγητές της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και για τα καλά λόγια με τα οποία αναφερθήκατε στις ε, υπηρεσίες του γραφείου μου. Νομίζω ότι τα θέματα είναι κοινά, είναι σημαντικά, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και ίσως είναι ε, συμπτωματικό που έγινε μια μέρα μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως ε, ε, γι' αυτό ακριβώς είχατε και πρόσφατη τη συζήτηση και θέλετε θίξατε το θέμα. Αναφερθήκατε στη διαφάνεια Αναφερθήκατε στη δυνατότητα switching, αλλαγής, φορέα και βεβαίως το σημαντικό να έχουν την γνώση οι, ε, οι πολίτες, οι καταναλωτές ότι έχουν δυνατότητα ε, αλλαγής παρόχου. Άρα καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά ε, το, την, την προσφορά Επίσης, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, ε, προσβασιμότητα ε, και ε, όροι εφαρμογής και περιορισμοί όσον αφορά τις διαδικασίες. Επίσης, οπωσδήποτε το θέμα των περιορισμών όσον αφορά τα τερματικά και τον εξοπλισμό των τερματικών. Βεβαίως, εσείς θα συζητήσετε το θέμα και θα πάρετε την τελική απόφαση, αλλά Βεβαίω, θα πρέπει να ξέρετε επί ποιων θεμάτων θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις και τι σημαίνει το ένα ή το άλλο πράγμα. Ε, το θέμα του switching είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα πρέπει να μπει και το θέμα των ε, αριθμών. Ε, και βεβαίως θα πρέπει η εφαρμογή του, της αλλαγής του, του φορέα να γίνεται από την πρώτη μέρα ε, και να μην υπάρχουν πολλοί περιορισμοί όσον αφορά τον χρόνο παραμονής ε, κτλ. Ε, το, το σημαντικό που λέμε πάντα είναι ε, να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ε, αποτρεπτικές διαδικασίες για την αλλαγή φορέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα επαγρυπνήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Για τον κύριο Ροσφόρ, βεβαίως λαμβάνω υπόψη του σοβαρά όλα αυτά τα οποία είπε. Ε, θα υπάρξει ο κώδικας αυτός για το 2012. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι ε, όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, εννοώ εμπιστοσύνη στις online αγορές ή συναλλαγές. Γιατί οι online συναλλαγές είναι πλέον κομμάτι με μεγάλο των συναλλαγών μας και της αγοράς. Ε, ε, ε, εμείς θέλουμε τα δικαιώματα να είναι ευνόητα, εύληπτα και οπωσδήποτε να γίνουν ευρύτατα γνωστά. λέμε ότι περισσότεροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν ακόμα ένα 27% Ευρωπαίων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο. Ε, θα πρέπει να τους πούμε ε, ότι πρέπει και αυτοί να μπουν στο διαδίκτυο γιατί χάνουν πολλά. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερωθούν επομένως για το τι σημαίνει, τι δυνατότητες τους ανοίγει το ε, διαδίκτυο και να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων. Τώρα, ο ε, οδηγός χρήσης ε, για το διαδίκτυο, για τους καταναλωτές, ε, θα τα εξηγεί όλα. Απαντώνται οι συχνότερες ερωτήσεις. Για τον κύριο Αρίας τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Χθες πραγματικά εντυπωσιάστηκα πριν ε, ακουστεί ότι θα υπάρξει και μια μεγάλη ε, πρωτοβουλία, ε, εντυπωσιάστηκα λέγω γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα έτσι ώστε να προωθηθούν οι φάκελοι σχετικοί με το ίντερνετ. Και πραγματικά το γεγονός ότι και οι G8 ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και με τις διαδικασίες αυτές ε, πραγματικά ε, καταδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Τα συζητούν σήμερα στην Τοβίλ. Και καταδεικνύεται σαφέστατα ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ένα θέμα το οποίο σαφέστατα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή με σαφήνεια, γιατί παίζει και μεγάλο ρόλο στη στρατηγική ε, του 2020. Χωρίς την ε, digital agenda δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ε, σύμφωνα και με αυτά που είπατε, στην ίδια τροχιά ε, αυτών που είπατε, δηλαδή ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με τρόπο ε, ρεαλιστικό Θα πρέπει να ξέρουμε ε, ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούμε να τη διευθετήσουμε. Ε, όχι απαραίτητα με καινούριου κανόνες και καινούριου νόμους κτλ. Να δούμε όμως κατάματα την κατάσταση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Μέρντοκ. Και αν δεν τα διαβάσετε, παρακαλώ να τα διαβάσετε. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και είναι πιο σημαντικό γιατί ε, αναφέρεται στην εκπαίδευση, αναφέρεται στη νέα γενιά, αναφέρεται στους νέους, ε, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Ε, και βεβαίως κύριε Πρόεδρε πρέπει να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι με όλα αυτά τα θέματα, είναι ε, στο πορτφόλιό μου, είναι στα θέματα που με απασχολούν. Αλλά ε, εδώ ε, υπάρχει μία αντιστροφή των συνήθων διαδικασιών. Εδώ αναφερόμαστε στους νέους που πρέπει να ξεκινήσουν και συνέχεια κατεβαίνει η ηλικία των ανθρώπων ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. 12χρονα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ήδη εντυπωσιάζονται από το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του. Επομένως θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και ε, όταν μιλάμε πλέον για εκπαίδευση θα πρέπει να αναφερόμαστε στα καινούργια εργαλεία, σε αυτά που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να μην χαλάμε, σπαταλάμε το χρόνο μας με πράγματα τα οποία δεν θα ενδιαφέρουν τα, αγόρια και τα, τα νεαρά αγόρια και τα νεαρά κορίτσια. γιατί ξέρετε ότι ε, στο facebook και στο twitter μιλάνε τα παιδιά, στο ebay πιο πολύ τα κορίτσια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τρία χρόνια πριν κανείς αν έλεγε ε, για το facebook ενδεχομένως να γελούσανε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν αλλάζουν σε σειρά ετών, αλλάζουν σε σειρά μηνών. Σε δύο-τρεις μήνες όπου έχουν αλλάξει τα πάντα. και επομένως ε, διαρκώς αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού και εμείς ε, πρέπει να ακολουθούμε, ε, η δημοκρατία αυτό είναι, να ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να προσαρμόζει βάζοντας όρια κτλ. Αλλά καμιά φορά χάνουμε και την μπάλα λίγο γιατί προχωράνε τόσο γρήγορα τα πράγματα αυτά που πραγματικά μερικές φορές χανόμαστε. Η σκηνή αλλάζει και πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να έχουμε τις αντένες μας ε, σε εγρήγορση γιατί αν χάσουμε την αγορά και τις εξελίξεις της αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Και εάν μπορούσαμε να επανέλθουμε στο θέμα της εκπαίδευσης ε, και εγώ δουλεύω πολύ και με την συνάδελφό μου την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου ε, και βεβαίως δεν είμαι εδώ για να σας υποδείξω ε, τη δικιά σας ημερήσια διάταξη με την πρέπει να ασχοληθείτε, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Κυρία Ράπτη. θα ελέγξει η Κομισιόν τους νέους κανόνες στην επόμενη βεβαίως ετήσια έρευνα. και είναι γεγονός ότι η Κομισιόν μπορεί να ε, πάρει διορθωτικά τεχνικά μέτρα για το 112. Όμως, ο εθνικός ε, ε, νομοθέτης είναι αυτός ο οποίος ε, θα πρέπει να ασχοληθεί με τα εθνικά κριτήρια. Ε, επομένως, μαζί και οι δύο πλευρές θα πρέπει να δουλέψουν. Για την ενίσα τώρα... Θα χρησιμοποιήσω ένα φαλτήριο την ερώτησή σας για να πω ότι και οι τρεις επίπροποι που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί καταφέραμε να ε, βάλουμε στο ίδιο τραπέζι διάφορους εμπλεκόμενους ε, φορείς. Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο μαζί ε, και με εμπειρογνώμονες ε, όχι μόνο δηλαδή τα τρία θεσμικά όργανα, ε, ασχολούμαστε ε, με την έρευνα αυτή. 1η Ιουνίου, πολύ κοντά δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η διαδικασία και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί μετά από πολλά χρόνια και από πολλή συζήτηση και το Συμβούλιο και η Κομισιόν είναι σε θέση να δώσει, να παραδώσει κατά κάποιο τρόπο ένα αποτέλεσμα και επομένως η ΕΝΙΣΑ, γιατί ξέρετε ότι η ΕΝΙΣΑ είναι ένα δίκτυο ας πούμε ε, που ασχολείται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου ε, και επομένως ε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα τόσο σοβαρά όσο είναι οι cyber attacks, αυτές οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αύριο έχουμε συμβούλιο και θα υπάρξει ενημέρωση για τα θέματα αυτά. Um, δεν θα μιλήσουμε για location, δεν, προτείνω, δεν προτείνουμε καμία αλλαγή, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, το θέμα της Ενίζα θα μας ε, απασχολήσει. Αναφέρομαι σε αυτήν την ε, την ε, οργάνωση, ας πούμε, τον οργανισμό της ΕΝΙΖΑ που βεβαίως θα πρέπει ε, να είναι σε θέση να δώσει ε, πληροφορίες και να βοηθήσει τη διασύνδεση των διαφόρων capitals. Οπωσδήποτε εμείς, πρωτεύουσαν, συγγνώμη, ε, και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι διασυνδέσεις να είναι σωστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι οι ερωτήσεις σας ε, είχαν ως αποτέλεσμα να ακούσουμε πολύ πλούσια παρουσίαση από την κυρία Ντεκρούς. Ε, δυστυχώς ε, ο επόμενος γύρος ερωτήσεων ε, θα είναι πάρα πολύ πιο σύντομος και οι απαντήσεις της κυρίας Επιτρόπου θα αναγκαστούν να είναι πιο σύντομες. Παρακαλώ όλοι όσοι θα λάβουν το λόγο πάρα πολύ σύντομα. Κυρία Βάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη παρόλο που θα ήθελα να ευχαριστήσω αναλυτικά την Επίτροπο της οποίας την εργασία εκτιμώ ιδιαίτερα. Το καταλάβατε φαντάζομαι. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, Αναφερθήκατε στην ασφάλεια στο κυβερνό χώρο. Από την άλλη μεριά αναφερθήκατε και στους νέους ε, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και την ε, δημιουργικότητά του σαν. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέοι χρησιμοποιούν αυτούς τις δυνατότητες πολλές φορές πολύ ελαφρά την καρδία και βλέπουμε ότι βρίσκονται συχνά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις όλο αυτό το mobbing, ε, δίωξη των, των, από τους άλλους φίλους τους στο διαδίκτυο είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ε, εφόσον υπάρχουν τόσο μεγάλα ατυχήματα ακόμα, είτε τα θέλουμε είτε δεν τα θέλουμε, ήταν προγραμματισμένα από κάποιους ή όχι, όσο γίνεται αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ προβληματικό να υπάρχουν στοιχεία υγείας ε, των ανθρώπων ε, στη, στο διαδίκτυο δεν είναι το ίδιο με το να έχουμε τα στοιχεία ότι κάποιος αγορέ κάποια παπούτσια. Το κύριο μου ερώτημα αφορά την πρωτοβουλία σας με τους άλλους συναδέλφους της Επιτροπής, φαντάζομαι, για τις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Ξέρω ότι και στη Γερμανία παντού ε, στην Ήπεθρο χρησιμοποιείται αυτό έντονα και χρησιμοποιούνται και πόροι των διαθροτικών ταμείων. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον έχουν απορροφηθεί όλα τα κονδύλια που διαθέτει η Επιτροπή. Θέλετε να αυξήσετε τον προπολογισμό γιατί υπάρχουν ορισμένες κοινότητες για τις οποίες είναι πάρα πολύ ε, προβληματικό να προσφέρουν για όλο το σύνολο της επικράτειας ε, εκεί ε, νέα συστήματα. Ο κύριος με ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι πολύ συναρπαστική, είναι μια πάρα πολύ θετική προοπτική. Καλό θα ήταν να έχουμε αυτές τις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες αλλά για να γίνει και να είναι και εφικτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία. Θα χρειαστεί να είναι εφικτό από πρακτικής πλευράς να μπορούν κάποιες επιχειρήσεις να παίρνουν πανευρωπαϊκές άδειες. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, τις προάλλες παρουσίασε ο Επίτροπος Μπαρνιέ τον οδικό χάρτη για την πνευματική διοκτησία. Για να είμαι απολύτω ειλικρινή, δεν βλέπω τις μεταρρυθμίσεις που θα ήταν απαραίτητε, ακόμη και για να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα θεμέλια για μια τέτοια νέα αγορά. Έχετε να σχολιάσετε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είμαι βέβαιο ότι έχει να σχολιάσει, λέει ο πρόεδρος. Τέλος, Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την εξαιρετική της παρουσίαση. Νομίζω κύριε Κρούσα σας ευχαριστώ εξ ονόματος όχι μόνο όλων των βουλευτών αλλά και όλων των Ευρωπαίων οι οποίοι μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. Η μείωση των τιμών περιαγωγής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό δεν είμαι βέβαια υπέρμαχος όλων όσων γίνονται στην αγορά, ε, αλλά προσπαθούμε να λειτουργήσει εύρυθμα η αγορά. Και χαίρομαι που επιχειρείτε κάτι καινούριο και ξέρω ότι στις 22 Ιουνίου θα δημοσιεύσετε ένα έγγραφο. Στα ΜΜΕ πάντως έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για κάποια εσανότατες τιμές ε, σε ό,τι αφορά την περιαγωγή. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. 24 cent θα είναι η μέγιστη τιμή το 2014 και 50 cent θα είναι η ανώτατη τιμή για το downloading πάλι το 2014. Και το cloud computing είναι κάτι το οποίο πράγματι εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς μέχρι το 2014. Μιλάμε για 35 δις ευρώ μέσω αυτού του cloud ε, computing. Καταπληκτικό θα ήταν κάτι τέτοιο, να περιορίσει δηλαδή η επιχείρηση το κόστος στην τεχνολογία των επικοινωνιών ή το κόστος της ενέργειας που μπορεί να μειωθεί. Βέβαια έχουμε και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινούν διαπραγματεύσεις με την ε, κοινή γνώμη, μάλλον διαβουλεύσεις με την κοινή γνώμη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να το σχολιάσετε, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις τελευταία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επιτρόπε, έχετε το λόγο. Ας ξεκινήσω με ένα ζήτημα που τόσο άλλος με απασχολεί ιδιαίτερα και το οποίο σχετίζεται με όλα όσα διακυβεύονται με αυτά τα οποία είπαμε δηλαδή θέση των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην προκειμένη περίπτωση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι η βάση της οικονομίας μας. Και όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας, για οικονομική ανάπτυξη, αυτή η κατηγορία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που είτε δημιουργούν είτε δεν δημιουργούν θέση άρα ανάλογα συμβάλλουν και στην οικονομία. Αυτό το οποίο συζητούμε λοιπόν έχει τη μεγάλη πρόκληση να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Όχι μόνο οι μεσαίες αλλά και οι μικρές. Και αυτό να γίνει διασυνοριακά. Για μένα το ιδανικό θα ήταν όχι να είναι πιο διαφανείς οι διαδικασίες, αλλά να υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση. Μιλάμε για ενιαία αγορά, αλλά όχι απλά για την ενιαία αγορά, μιλάμε για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Και έχουμε να κάνουμε πολλά και στα δύο μέτωπα. Για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία συμφωνώ. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε. Συλλογική είναι η απόφαση, η δική μου θέση είναι σαφή. Σαφής. Αυτό το οποίο πιέζω είναι να μην σταματήσει με τις διαβουλεύσεις ή με την πράσινη βίβλο, αλλά να ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Οι προκλήσεις είναι συναρπαστικέ και επανέρχομαι στην χθεσινή μέρα και στι προηγούμενε ημέρε. Με αυτή την αλλαγή η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική. Και επειδή μιλάμε για τις προκλήσεις και με βάση τις χθεσινές μας εμπειρίες θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προκλήσεις για αύριο, για το μέλλον. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοξίας. Να μην παρεξηγήσετε. Νομίζω ότι όλοι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες χρειάζεται να αμείβονται αξιοπρεπώς και πρέπει αυτό να το προστατεύσουμε. όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού γενικώ. Αν όμως δεν δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να λαμβάνουμε υπόψη και το σήμερα αλλά και το αύριο, τότε θα κάνουμε ένα λάθος. Θα έχουμε περιμείνει πάρα πολύ και θα έχουμε χάσει χρόνο. Δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, έτσι μιλάω και για τα δεδομένα Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, ε, ε, βρίσκουν το δρόμο τους μέσα από παράνομα κυκλώματα. Πολλές φορές δεν το κάνουν ε, σκοπίμως, γιατί είναι υπέρ της παρανομίας, αλλά γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο πολλές φορές. Και αν μου επιτρέπετε. Μην κάνουμε σφαλμένη κρίση όμως ότι είναι μόνο νέοι. Δεν είναι μόνο νέοι αυτοί. Λοιπόν, Τούτου λεχθέντος έχουμε τεράστιο περιεχόμενο, τεράστιο πλήθος περιεχομένου το οποίο παρέχεται. Στην Όπο Ανατολή παράγεται τεράστια ποσότητα αγαθών, αλλά και καινοτομία ενώ στην ε, αποδύση θα έλεγα, το περιεχόμενο είναι αυτό στο οποίο αριστεύουν. Εμείς αγοράζουμε και από τους μεν και από τους δε τελικά. Αλλά δεν μπορούμε. Πρέπει να έχουμε και εμείς μια δική μας αγορά, τις δικές μας επιχειρήσεις. Πρέπει να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας σε, αυτή την παγκόσμια, σε αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις. Γι' αυτό οι επενδύσει είναι τόσο σημαντικέ, παραδείγματο χάρη στην ευρυζωνικότητα. Γι' αυτό μιλάμε για όλο αυτό το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε συστήματα, αλλά επικαιροποιημένα. Και χρειαζόμαστε και την υποδομή για την ανάπτυξη δεδομένων. Πραγματικά είναι τρομερό. Και όπως γνωρίζετε, το Μάρτιο διοργάνωσα μία συνάντηση με τους ε, εκτελεστικούς διευθυντές όλων όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό και τηλεπικοινωνίες αλλά και μετάδοση, φορείς μετάδοσης, ε, βιομηχανία κτλ. Είπα δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας γιατί εσείς έχετε τις δικές σας ευθύνες και πρέπει να αποφασίσετε αλλά θα πρέπει να υιοθετήσετε μια δημιουργική προσέγγιση να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και να σκεφτείτε νέα μοντέλα, νέα επιχειρηματικά, επιχειρησιακά μοντέλα. Και βέβαια για μένα πολύ σημαντικό είναι το θέμα των επενδύσεων, ας πούμε, όταν μιλάμε για την ευρυζωνικότητα. Δεν ξέρω, μιλάμε για 270 δις ή 250. Δεν είναι χαρτζηλίκι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει κέρδος, κανείς δεν στοιχηματίζει τα λεφτά του. Αυτό είναι το καταπιταλιστικό σύστημα. Αυτό λοιπόν το οποίο εδώ διακυβεύεται είναι ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να βάλουν το περιεχόμενο στους αγωγούς στο δίκτυο πρέπει να έχουν και τις ευκαιρίες. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Εγώ είμαι βέβαιη ότι χρειάζεται ε, περισσότερο, κάτι περισσότερο από την απλή εκπόνηση πράσινης βίβλου. Για το cloud computing το είπαμε. Για την περιαγωγή, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω αν τα αριθμητικά στοιχεία που μου αναφέρατε είναι ακριβή, αλλά σύντομα θα επανέλθω. Με το cloud computing συμφωνώ απόλυτα ότι η προστασία των δεδομένων είναι ένα must. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον το cloud computing και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή θα πρέπει να το δούμε ε, σε όλο το κλάδο. Για τα ορφανά έργα, για το οπτικοακουστικό <clears throat> τομέα, θα έχετε νέες προτάσεις, το υπόσχομα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας, το είπα αυτό. Διαρθρωτικά ταμεία. για τις επενδύσεις. Τα διεθντικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής υπάρχουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Χθε όμως αποφασίστηκε ένα νέο ταμείο. Είχαμε ένα μίνι σεμινάριο του Σώματος των Επιτρόπων, αλλά θα το συζητήσουμε στην επίσημη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων για να έχουμε τη χρηματοδότηση ε, για την υποδομή, υποδομή ενέργειας και ευρυζωνικότητα ICT τεχνολογίε πληροφοριών και επικοινωνιών. Και εκεί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και σαρπαστικό θέμα. Άσκηση μόχλευσης. Αν εμεί μπορούμε να βάλουμε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι, τότε με τις τράπεζες και αν έχουμε μια κοινή αντίληψη και θεώρηση των ευκαιριών μπορούμε να προχωρήσουμε. Νέοι, νεολαία και ασφάλεια του κυβερνοχώρου πράγματι είναι ένα από τα θέματα για τα οποία η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι και τα πιο ευάλωτα άτομα και αυτούς έχουμε στο επίκεντρο των ε, προσεγγίσεών μας. Χρειαζόμαστε τους γονείς, χρειαζόμαστε επίσης ενημέρωση προς τους νέους. Προσοχή όταν πατάτε το κουμπί send, αποστολή. Αναλαμβάνετε κινδύνους. Αλλά και τους γονείς πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε. Και έρχομαι στο πρώτο μου σημείο, κύριε Πρόεδρε. Κάποιες φορές οι νέοι πράγματι είναι πιο μπροστά σε σχέση με τους γονείς. Άρα θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι γονείς στις νέες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα με τους νέους, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να κάνουν τα δικά τους, γιατί πραγματικά μιλάμε για πολύ ε, μεγάλο θέμα αυτό της κυβερνοασφάλειας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί δεν απαντήσατε απλώς στις ερωτήσεις, αλλά κάνατε παρουσιάσεις, αναφερθήκατε σε στοιχεία καινούρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας, ευχαριστούμε πολύ, ε, ευχαριστούμε και τους διερμηνείς και ευχαριστούμε τον πρόεδρο οι διερμηνείς. Επόμενη συνάντηση, 14 Ιουνίου, 3 το απόγευμα και 15 και 16 επίσης θα συνεχίσουμε. Θα τα πούμε τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας.